Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε αμέσω. Έχουμε ήδη καθυστερήσει λίγο. Θα ήθελα να σα ε, ζητήσω να περάσουμε απευθεία στην έγκριση τη ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχουν ενστάσει και θα ήθελα να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 28 η Νοεμβρίου και της 3 η Δεκεμβρίου. Παρακαλώ. Μία πρόταση. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ναι. Θα ήθελα να συζητήσουμε και τη βουλγαρική περίπτωση και αν δεν γίνει αυτό σήμερα, τότε τότε αποσιοποιητικά. Okay? It's possible. Okay. Уважаема госпожо председател, Πρόεδρε, επαναλαμβάνω η διαφθορά στη Βουλγαρία αυξάνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα και θα ήθελα να τεθεί ένα θέμα για τη συζήτηση της διαφθοράς στη Βουλγαρία και αν αυτό δεν γίνει σήμερα τότε θα γίνουν τα πράγματα πολύ άσκημα στη Βουλγαρία γιατί ξέρετε ότι έγινε μια απόπειρα πρόσφατα. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα, τότε να το συζητήσουμε όπο, όσο γρηγορότερα γίνεται. Σας ευχαριστώ και ελπίζω η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών να επιδειχθεί και η Ένωση να μην αρνηθεί να συζητήσει τέτοιες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε σήμερα στη συνεδρίαση των συντονιστών. Δεκτό λοιπόν το αίτημά σα και θα προταθεί στη συνεδρία των συντονιστών. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά και την ημερήσια διάταξη, έχουμε μία αλλαγή. Στο σημείο 4 προβλεπόταν η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Ε, αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Σας ζητώ λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με την αλλαγή αυτή. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε τα πρακτικά από τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, τις 28 Νοεμβρίου και τις 3 Δεκεμβρίου, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Σημείο 3 τώρα, δύο ανακοινώσεις. Ο κύριος ε, Σαλντεμπίνεφ που προέρχεται από τη Βουλγαρία είναι πλέον μέλος της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Ε, από την Ευρώπη της Ελευθερίας και Δημοκρατίας και ο Γιάνν Φιλιπ Άλμπρεκτ γίνεται ο νέος συντονιστής των Πρασίνων ε, αντικαθιστώντας τον Μπαρτ Στάις. Όπως ε, γνωρίζετε η συνεδρίαση αναμεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Europal TV και σήμερα θα γίνει το απόγευμα η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών των συντονιστών από τις 5.30 και μετά. Πέμπτον, όπως γνωρίζετε, η εντολή της Επιτροπής μας προβλέπει την ε, ε, παρουσίαση μιας ενδιάμεσης έκθεσης και μιας τελικής έκθεσης του εισηγητή, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι θα παρουσιάσει κάποια ε, στοιχεία σε τρία έγγραφα εργασίας για τις αρμοδιότητες της δουλειά μας, για το οργανωμένο έγγραμμα, τη διαφθορά και την... Ε, ανακύκλωση χρήματος. Σήμερα ο κύριος Γιακολίνο θα ήθελε να παρουσιάσει το δεύτερο έγγραφο εργασίας. και βάσει των διαφόρων παρουσιάσεων των εμπειρογνωμόνων ε, στις ε, δημόσιες ακροάσεις της Επιτροπής μας ε, καταρτίστηκε και αυτή η έκθεση. Θα πρόκειται λοιπόν για μία σύνοψη τη συνεισφορά των συναδέλφων αλλά και τη συνεισφορά που είχαμε από τις δημόσιες ακροάσεις που είχαν ως θέμα τη διαφθορά. Η συζήτηση θα γίνει ως εξής. 20 λεπτά θα έχει ο κύριος Γιακολίνο για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Από εκεί και πέρα δύο λεπτά στον κάθε προβουλευτή που θα ζητήσει το λόγο, με προτεραιότητα φυσικά στου συντονιστέ, και κατόπιν θα απαντήσει ο εισηγητή. Παρακαλώ κύριε Κολίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για την πολύ ουσιαστική συνεισφορά τους σε αυτό το έγγραφο εργασίας, το οποίο καταρτίστηκε χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη και της γραμματείας Συζητήσαμε τα θέματα που αφορούν το οργανωμένο έγκλαμα στο πρώτο έγγραφο εργασία και κατόπιν κάναμε μία απόπειρα να βρούμε λύσεις τις οποίες θεωρούμε ότι συνάδουν και με το πνεύμα της εντολής ε, που έχει ε, δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ετοιμάσαμε ένα έγγραφο εργασίας που προσπαθεί σε 16 σελίδες να συγκεντρώσει τη συνασφορά και των θεματικών εγγράφων τα οποία ε, έδωσαν οι συνάδελφοι Γκάμπριελ Γουάιρλεν, Γκίγιον και Σκυλακάκης. Όλες ε, πολύ εύστοχες συνεισφορές, ε, πολύ σημαντική η υποστήριξή τους και φυσικά όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο έγγραφο. Ο κύριος Ντεγιόγκ ασχολήθηκε με τη διαφθορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μετά ασχολήθηκε με τη διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Γκάμπριλας ασχολήθηκε με τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις. Ε, ο κύριος Κυλακάκης με τη συστημική διαφθορά στη δημόσια διοίκηση στα κράτη-μέλη και ε, κάποια μέτρα για να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυρία Βάιλερ στη χρήση των ευρωπαϊκών κοντήλιων από πλευράς οργανωμένου εγκλήματος. Έγιναν ε, πολύ ενδιαφέρουσε ακροασει, ήταν πολύ συνεχή η εργασία μας και από τι ακροασει είδαμε και τι διαστάσει ενό φαινομένου που έχει διεθνής, ε, διεθνή επιρροή και δεν είναι απλώς ευρωπαϊκό. Θα σας πω τα πιο σημαντικά στοιχεία κατά την άποψή μας ε, με τα, βάση τα όσα κάναμε όλοι μαζί από κοινού και θα ήθελα να τα συνοψίσω για τους ε, συναδέλφου και για όσου μα ακούν. Στόχος είναι να έχουμε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, κοινά νομικά πρότυπα, δείκτες για να μπορέσουμε να μετρήσουμε αυτά τα φαινόμενα, προληπτικά μέτρα προκειμένου να μειώσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι ενδυμικό και είναι παρόν σε πολλά κράτη-μέλη με πολύ υψηλά ποσοστά μεγαλύτερη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση που θα συνδέεται φυσικά και με μια μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης ε, προώθηση της νοοτροπίας της ανάληψης ευθύνης των ηθινόντων, των πολιτικών, ε, μέρημνα για τους ε, ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται και ε, δίνουν πληροφορίες στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Έχουμε προβλέψει επίσης και αυστηρά μέτρα ενώπιον των πολιτικών, οι οποίοι αμάυρωσαν τη δραστηριότητά τους με ε, συμπεριφορές οι οποίες ε, δεν συνάδουν φυσικά με το έργο τους και είναι δευτερμένοι, προβλέπονται και προληπτικά μέτρα. και προβλέπεται να μην ε, υπάρχει δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν ε, διοικητικά ή κυβερνητικά καθήκοντα. Ε, δίνουμε και κάποιες σημαντικές ενδείξεις για τα κόμματα, για την κατάρτιση του κώδικα διοντολογίας τους, καθώς επίσης ένα κώδικα διοντολογίας για τις επιχειρήσεις, ένα μητρό για τις ομάδες πίεσης, λευκές λίστες επιχειρήσεις για να δίνεται πιστοποίηση με τη δημόσια διοίκηση. Προβλέπεται επίση και ανταλλαγή κάποιων πληροφοριών, όπω για παράδειγμα στην Ιταλία, το τι γίνεται με τι ανταλλαγέ χρημάτων. Και θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει και διάφορα άλλα πλεονεκτήματα ε, και να εξετάζονται και άλλοι πόροι, όχι μόνο υλικά αγαθά. Επίσης μας ενδιαφέρει να γίνονται σε σύντομο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί το κράτος και το δικαίωμα και την εξουσία να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να παραγράφεται το αδίκημα. Να έχουμε δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο θα γίνεται ανα ε, βαθμούς ε, δικαιοδοσίας και από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταδικαστεί ε, δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιες ε, ε, προσφορές σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Παραδείγματο χάρη, αν μια επιχείρηση που έχει καταδικαστεί στην Ιταλία και υπάρχει ποινή, δεν θα μπορεί η επιχείρηση αυτή να δραστηριοποιηθεί και σε άλλα κράτη-μέλη και για λόγους αμοιβαιότητας το ίδιο θα συμβεί και αν η ποινή αυτή έχει εκδοθεί ε, για μια επιχείρηση στην Ιταλία που δεν είναι Ιταλική ή σε κάποια άλλη χώρα μέλος με τις ίδιες διαδικασίες. Να υπάρχει δυνατότητα ε, επίσης ανιχνευσιμότητας ε, των οικονομικών ροών, να υπάρχει κατάρτιση των δικαστικών η οποία να είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι ήταν μέχρι τούδε και επίσης να υπάρχει συνεργασία. Ορισμένες φορές είναι ε, διασυνοριακά αυτά τα δικήματα, επομένως χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, με τη Europol, με τη Eurojust, την Olaf και φυσικά και με τρίτες χώρες. Ε, μεγαλύτερη συνεργασία με, την, ε, τον ΟΗΕ, τον ΟΣΑ, συμμετοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κρέκο και επίσης να υπάρχει δυνατότητα να κυρώνονται και να ε, προσυπογράφουμε όλες αυτές οι συμβάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν ιστηρή στήριξη στην ε, αντιμετώπιση της διαφθοράς. Να ενισχύσουμε τις κοινέ ομάδες έρευνας και να δώσουμε και ε, ένα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μπορεί να εκδώσει ποινές σε τέτοιες ε, σε τέτοια δικήματα τα οποία είναι διεθνού φύσεως. Ε, στις τελευταίες ημέρε συναντήθηκα και με τους κοιόδης συζητητέ και συζητήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας ανέφερα προσπαθώντας να βρούμε κοινό σημείο και ε, χάρηκα ιδιαίτερα διότι υπάρχουν κοινά σημεία επαφή και τους ευχαριστώ ιδιαίτερως για την διαθεσιμότητά τους και τη γενεοδορία τους στα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Ο κύριος Κίλκοφ ε, πρότεινε να λάβουμε υπόψη και κάποιες βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο θέμα ε, των ε, κονδυλίων αλλά και στις κατοχώρες και να δοθούν περισσότεροι πόροι στη Europol και στην Όλαφ και να δούμε για ποιο λόγο η σύμβαση του ΟΣΑ για την ε, διαφθορά των δημοσίων λειτουργών ε, δεν έχει ακόμα κυρωθεί σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση και είμαι πεπισμένος ότι από εκεί και πέρα θα ενημερωθούμε Ο κύριος Κυλακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει καλύτερη κατάρτιση και να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, στα στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και να δοθεί και κάποιος χώρος στις αυτόνομες πρωτοβουλίες ε, που αναλαμβάνουν οι αρχές ώστε να μπορούν να ε, κάνουν το έργο τους. Ο κύριος Ταβάρες ασχολήθηκε κατά βάση με το δημοσιογραφία και την έρευνα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, τι μελιγενέστε. Ε, τα επόμενα βήματα ε, σε κάποιο βαθμό τα έχει υπογραμμίσει και η Πρόεδρος. Θα περάσουμε δηλαδή στην παρουσίαση του τρίτου εγγράφου για την ε, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, ε, στο οποίο μαζί με τη Γραμματεία και με τους συναδέλφους που ετοίμασαν τις δύο εκθέσεις Υπολογίζουμε τις επόμενες εβδομάδες, στις 18 Φεβρουαρίου, να σας παρουσιάσουμε το έγγραφο για την ομοιοποίηση παρανόμων εσόδων, ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την παρουσίαση της ενδιάμεσης έκθεσης. Τώρα, αυτό το έγγραφο είναι, ακόμα, είναι σε προχωρημένο στάδιο και φυσικά θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμε οι συνεισφορές ε, των συναδέλφων Ποργέτσιο και Ταβάρες ε, για την ενδιάμεση έκθεση θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα χρήσιμα στοιχεία τα οποία είχαμε και από τις ακροάσεις μας ε, και ε, τις επισκέψεις των αντιπροσωπιών που μας βοήθησαν να διελευκάνουμε ε, κάποια πράγματα και αυτή που θα κάνουμε τον επόμενο μήνα. Και την προηγούμενη εβδομάδα ζητήσαμε από τις πολιτικές ομάδες να μας δώσουν ένα κατάλογο των προτεραιοτήτων τους ε, βάσει των οποίων θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια πώς θα ολοκληρώσουμε την έκθεση εντός και του χρονοδιαγράμματος με βάση την εντολή που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν σίγουρα χρήσιμη η εμπειρία κάποιων ε, εθνικών ε, νομοθεσιών. Ε, να δώσω για παράδειγμα της Δανίας, διότι ήταν πολύ επικοδημητική ε, το τι γίνεται στη χώρα αυτή μεταξύ κυβέρνησης και ελεγκτικού συνεδρίου. Πρόκειται για μια σημαντική ε, πληροφορία, διότι το τι κάνει το ελεκτικό συνέδριο ε, είναι συγκεκριμένες ενδείξεις και η κυβέρνηση υποχρεούται να τις λάβει υπόψη της για να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη λύση και συγκεκριμένη γνώμη για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ακόμα και τι συμβαίνει σε κάποια άλλα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τη στήριξη της Eurojust με την προοπτική και μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία που θα ασχολείται με συγκεκριμένα δικήματα, όπως για παράδειγμα τη διεθνή διαφθορά. Ε, ελπίζουμε ότι θα συμπεριληφθεί και αυτή σε αυτά τα θέματα και ασχολήθηκαμε και θα ασχοληθούμε εν συνεχεία πάντα με επικοδομητικό πνεύμα με τους ελέγχους για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, ιδίως ε, των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την πολιτική συνοχή στι περιφέρειε με στόχο τη σύγκληση και τέλος θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, προστασία για το δημόσιο λειτουργό ο οποίος ε, καταγγέλει παράνομες δραστηριότητες τις οποίες έχει διαπιστώσει στο χώρο εργασίας του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσει να λάβει δεόντως υπόψη όλες τις ε, πολιτικές κατευθύνσεις που θα δώσει η έκθεσή μας στο τέλος της θητείας. Και θεώρησα όμως ότι πρέπει πριν περάσουμε στο συμπέρασμα ε, να υπενθυμίσω στα πλαίσια του χρόνου και μου έχει δώσει η πρόεδρος, ότι το θέμα της διαφθορά είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με μια θεμελιώδη έννοια, την έννοια της ευθύνη. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να υπάρχει ε, σαφής ορισμός και σαφή, απλή, ευέλικτοι κανόνες, του οποίους μπορούμε να εφαρμόσουμε εύκολα. θα πρέπει να γίνει μια γενική προσπάθεια για να μετρήσουμε τη διαφθορά από όλους μας και η μέτρηση της διαφοράς ε, περιλαμβάνεται και σε κάποιες ταξινομήσεις που γνωρίζουμε και σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι ε, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ολοκληρώνοντας ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους πολιτικούς, τους δημοσίους λειτουργούς και όλους όσους έχουν ένα δημόσιο αξίωμα επιτάσσει να δοθούν σαφείς κανόνες, τουλάχιστον από δεοντολογικής ε, πλευράς και αυτό θα πρέπει να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να καθορίσει μια σειρά από κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν έμπνευση για να είναι διατάξει από εκεί και πέρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, και εμείς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να δώσουμε στη συνέχεια πολιτικές κατευθύνσεις και πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες θα κληθούν τα κράτη-μέλη από εκεί και πέρα να ε, ε, περάσουν στην νομοθεσία τους και να ε, αναλάβουν την ευθύνη για αυτές. Ολοκληρώνω λοιπόν, ε, δεν θα αξιοποιήσω όλο το χρόνο που μου έδωσε η Πρόεδρος και να υπενθυμίσω ότι στον κατάλογο των προτεραιοτήτων που έχουμε επισημάνει υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών με την ευρύτερη άνοια και να γνωρίσουν τι ακριβώς γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη, διότι είναι απαραίτητη αυτή η εμπειρία προκειμένου να γνωρίζουν τι συμβαίνει όπως γίνεται και με την, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, διεθνούς διαφθοράς, είπαμε ήδη ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί στο επίκεντρο ε, το όργανο αυτό το οποίο προβλέπεται από τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα είναι το μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει να συντονιστούμε και για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα είναι από τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε περισσότερο και εδώ η Επιτροπή αυτή θα έχει και τη δυνατότητα να ε, δώσει πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις. Και φυσικά όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στο τελικό έγγραφο και στο έγγραφο το οποίο θα παρουσιάσουμε στην ενδιάμεση έκθεση και στο τελικό το οποίο θα ετοιμάσουμε αφού εγκριθεί η ενδιάμεση έκθεση από το Κοινοβούλιο. Θα σταματήσω εδώ, εντός των χρονικών ορίων, γιατί θα ήθελα να ακούσω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ιακολίνο. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους και τους κοιόδης εισηγητές που συνεργάστηκαν για να ε, ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση και θα ήθελα να σας πω ότι ναι μεν υπάρχει ανάγκη μια θέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για το πώς θα αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα και εδώ δεν θα ήθελα να υπάρχουν παρανοήσεις. Πρέπει να ενισχύσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των Ευρωπαίων πελιτών. Και σε αυτό έχουμε ήδη καθυστερήσει, διότι η διαφάνεια είναι το μοναδικό αντίδοτο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, διότι όπως είδαμε συνεχίζεται, συνεχίζεται όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση αλλά και ε, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είδαμε τι έγινε στο τραπεζικό τομέα, διότι στις ε, δημόσιες ακροάσεις είχαμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε πώς ε, συγκεκριμένες συμπεριφορές ε, αντιμετωπίζονται παντού και τι ζημίες υπήρχαν ε, και τις διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να σας πω ότι κατά την άποψή μου η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ χαμηλή. Κανονικά πρέπει να κάνουμε μια νέα αξιολόγηση γιατί αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι ελάχιστα. Εσείς προηγουμένως αναφερθήκατε και στη δέσμη μέτρων που πέρασε στην Ιταλία στις 31 Οκτωβρίου. Πρόκειται όμως για ένα ε, ε, ε, πακέτο ελιπές, διότι δεν υπάρχουν όλα όσα θα έπρεπε να υπάρχουν. Και θα ήθελα να πω το εξής. Εμείς έχουμε καθήκον όπως εποπτεύουμε όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τις, ε, να εποπτεύσουμε και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε μια καλύτερη σύνθεση των όλων θεμάτων και να παρουσιάσουμε ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρό. Υπενθυμίσατε και δικαίως την ανάγκη να υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένοι κανόνες, ε, να υπάρχουν λευκές λίστες, να μην υπάρχει δυνατότητα να υποβάλει κάποιος υποψηφιότητα, να έχει καταδικαστεί. Και αυτό είναι θεμελιώδες, όχι μόνο ε, διότι είναι το σωστό, αλλά γιατί πλέον είναι πάγια πρακτική πολιτικών και συναδέλφων που έχουν καταδικαστεί επανειλημμένων και παρόλα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν δημόσια αξιώματα και στην κυβέρνηση και στις περιφερειακές κυβερνήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή έχουμε και πάλι προεκλογική εκστρατεία. Εγώ διάβασα, δεν ξέρω αν το διαβάσετε κι εσείς στον τύπο, κάποιες ε, πληροφορίες οι οποίες ε, κατά την άποψή μου αποτελούν ενδείξεις. Διάβασα για κάποιους υποψηφίους που έχουν απάντησαν ευγενικά στους δημοσιογράφους που τους ρώτησαν πώς και κάνετε υποψηφιότητα. Η απάντηση ήταν «Ε, εγώ πλήρωσα την προεκλογική εξαιρετία του ΤΑΔΕ, οπότε είναι πολύ λογικό να με συμπεριλάβει στη λίστα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ε, ισχυρά μέτρα ο λευκός κατάλογος αυτός της επιχειρήσης είναι σημαντικός για να μην επιτρέπεται να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είτε στη χώρα μας είτε σε άλλη χώρα ε, να έχουν καταδικαστεί και να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες. Και επίσης είναι σημαντικός ο ρόλος των μαρτύρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, είναι πολύ σημαντικό. Χρήζουν προστασία σε αυτοί οι άνθρωποι και θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους και τώρα να σας δώσω το λόγο και θα έπρεπε πριν ολοκληρώσω να σταθώ και στην ε, εφαρμογή των, του κώδικα δεοντολογίας των πολιτικών κομμάτων, γιατί εκεί διακυβεύεται όλο το παιχνίδι. Αν τα πολιτικά κόμματα δεν αντιληφθούν ότι πρώτα αυτά πριν ε, υπάρξει ευρωπαϊκός νόμος θα πρέπει να έχουν ένα κωδικό, ε, κώδικα δεοντολογίας στο κόμμα τους που θα ρυθμίζει συγκεκριμένες συμπεριφορές ε, και παρουσίες στους κόλπους του κόμματός τους. Να δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστέ. Έχει ζητήσει το λόγο ενώματος των φιλελευθέρων ο κύριος Νιούτον Ντάν. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Σαλβατόρε, πολύ καλό έγγραφο, ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι πλησιάζουμε στα τέλη Ιανουαρίου και έχουμε και άλλα δύο έγγραφα του Σαλβατόρε που προβλέπονται. Τα αναμένουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Τώρα συγκεκριμένα σχόλια για το έγγραφο αυτό για τη διαφθορά. Θα ήταν νομίζω καλό σε μερικά μέρη να γίνεται κάποια αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα. Μπορώ αν θέλετε να σας στείλω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συγκεκριμένες αναφορές που να λένε από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες για να μπορούν και οι άλλοι να τις επαληθεύσουν. Αυτό όμως είναι λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι ότι στην αρχή της έκθεσης του γίνεται ένας ορισμός της διαφουθοράς και θα ήθελα να συμπεριληφθεί εκεί η λέξη μυστικά και καλυμμένος γιατί αν θέλουμε διαφάνεια δεν θα υπάρχει. Αν υπάρχει διαφάνεια δεν υπάρχει διαφθορά. Λοιπόν θα έλεγα ότι στον ορισμό της διαφθοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κάπου η έκφραση ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ότι όλα αυτά γίνονται και καλυμμένα. Έπειτα, προβοκάτορες. Αυτά μου φαίνονται ύποπτα και περίεργα πράγματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μυστικούς προβοκάτορες. Άλλο. Στην τελική σύσταση ίσως πρέπει να πούμε ότι σε οποιαδήποτε οργάνωση η διαφθορά αρχίζει από το κεφάλι όπως βρωμάει το ψάρι δηλαδή. Ο Μάρτιν Σούλτς είναι εξαιρετικός πρόεδρος αλλά εάν υποθέσουμε ότι ήταν διεφθαρμένος, τότε και όλοι εμείς θα καταλήγαμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να γίνει εκεί να δοθεί κάποια εξήγηση ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ο συνάδελφος από τη Βουλγαρία μας μίλησε για τη διαφθορά εκεί. Σκεφτείτε από την άλλη μεριά τον κύριο Μπερλουσκόνη. Αν μια χώρα κατευθύνεται από κάποιον διεφθαρμένο είναι τρομερή καταστροφή και πριν από 100 χρόνια είχε υποθεί ότι όλη η εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Μάλλον δεν μπορούν να το μεταφράσουν αυτό οι διερμηνείς γιατί είναι τόσο δύσκολο, δύσκολη έννοια. Αλλά εννοώ απλώς ότι πρέπει από την ηγεσία να, υπάρχει, να αρχίζει η διαφάνεια. Νομίζω ότι πρέπει η Θεσμική Επιτροπή για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών κομμάτων να σκεφτεί το ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά στη χρηματοδότηση των κομμάτων και στη χώρα μου. Δεν ξέρω ούτε το δικό μου κόμμα πώς χρηματοδοτείται και ίσως να μην θέλω και να μάθω. Είναι τρομερά πράγματα αυτά. Ή δέστε τι κάνουν οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκράτες στην Αμερική που μαζεύουν εκατομμύρια δολάρια για τις εκστρατείες. Κάτι συμβαίνει εκεί. Και τέλος προ τα τέλη της έκθεσης όπου μιλάει για το ΙΤΑΒ τη χώρα μου είναι πολύ ευγενής ο Σαλβατόρε. Δεν νομίζω ότι όλα όσα λέει εκεί για την, το Ηνωμένο Βασίλειο αληθεύουν. Απλώς είναι πολύ ευγενής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμποργέτσιο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Δεν θα πω πολλά για την έκθεση, διότι νομίζω ότι το έγγραφο τα λέει όλα από μόνα του. Μια εξαιρετική και δύσκολο να την καταφέρει κάποιος σύνοψη των προβλημάτων που προκαλεί διαφθορά. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Ιακολίνο, διότι καταφέρετε με τη βοήθεια των συναδέλφων ε, που συνεργάστηκαν μαζί σας να μας δώσετε ένα πλήρες πλαίσιο του θέματος και επομένως ένα εξαιρετικό εφαλτήριο που αποτελεί σημαντικό βοήθημα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για να πούμε και του στραβού το δίκιο μέχρι τώρα δεν έχει κάνει και ό,τι μπορεί για τη διαφθάνεια και ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο ε, προκύπτει στην αξιολόγηση των θεμάτων αυτών και αυτό είναι η χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Ως Ιταλός, ε, τουλάχιστον όσον αφορά την ταυτότητά μου, Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος ε, για το θέμα αυτό, διότι ε, είχαμε συναρπαστικά γεγονότα. Θυμάστε άλλωστε την χρηματοδότηση η οποία ευτυχώς ε, σταμάτησε πάνω των 25.000 ευρώ στον αδερφό του, του Τολίνα, ο οποίος είναι ο νονός της Ιταλικής μαφίας αυτή τη στιγμή. Και πρόκειται για μια χρηματοδότηση η οποία ε, δόθηκε επιπλέον της χρηματοδόθηκε που δόθηκε στον Γκαετάνο Λίνα, ο οποίος ε, ήταν και ε, υπόδικος και τον ερευνούσε η αστυνομία, επομένω δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Να, να χρηματοδοτηθεί. Και το όνομά του φυσικά ήταν γνωστό της Πάση. Γι' αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν όσοι κάνουν προληπτικό έργο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προτείνω στον συνάδελφο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όμως, αλλά να προσέξει και αυτό και να επικεντρωθεί, αν γίνεται, λίγο περισσότερο στο θέμα της πρόληψης και του ελέγχου. Ε, βεβαίως, τα όσα λέγονται στο έγγραφο για την σημασία ε, της ε, αποτελεσματικότητας αυτού του προγράμματος Καπάτσι είναι ε, βασικά, αλλά το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως ένα στοιχείο που ε, επισημαίνει μια ανησυχία αλλά δεν προσφέρει τη λύση. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο το θέμα αυτό και ίσως θα έπρεπε να ε, εξετάσουμε και το ενδεχόμενο ενός μόνιμου παρατηρητηρίου το οποίο θα ε, περιλαμβάνει πρωτίστως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι αδιανόητο τόσο σοβαρά σφάλματα και αυτό το οποίο σας ανέφερα είναι απλώς ενδεικτικό παράδειγμα να συμβαίνουν χωρίς να υπάρχουν και ε, συνάφειες στις Βρυξέλλες, ε, στους υψηλά εσταμένους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όσον αφορά τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο ανέφερε και η Πρόεδρος και το ανέφερε και ο συνάδελφος από τους φιλελευθέρους, ε, θεωρώ ότι και αυτό είναι ουσιαστικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, διότι και αυτά έχουν καθοριστικό ρόλο στη σχέση μεταξύ ε, πολιτικής επιχειρήσεων, πολιτική επιχειρήσης εγκληματικότητα, πολιτική επιχειρήσης εγκληματικότητα μαφία. Και φυσικά αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εμείς ε, έχουμε την πρόσφατη εμπειρία που έφερε στο φως ε, γεγονότα πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να πω, εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά τα γνωρίζουμε. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, Ε, το τι γίνεται στη διοίκηση των κομμάτων ε, είναι πάρα πολύ ασαφές, ε, ακόμα και στις, στα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή. Υπάρχει αυτή η έννοια της αυτονομίας του Κοινοβουλίου και στην πραγματικότητα διαπιστώσαμε ότι κανείς δεν ελέγχει, κανείς δεν προσέχει, κανείς δεν είναι υπεύθυνος. Επομένως υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι απόλυτα φαιός και δεν αναλαμβάνει κανείς ευθύνες. Και αυτό είναι και το πιο σοβαρό. Κύριε Μποργέτζιο, αν γίνεται να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος. Και τέλος πάντων αυτό είναι συνήθως πρακτική, λέει ο κύριος Μποργέτζιο, και θα πρέπει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για το θέμα αυτό, να κάνουμε συγκεκριμένε προτάσεις και για τη χώρα μας τουλάχιστον υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα βάσει του οποίου τα πολιτικά κόμματα είναι μη αναγνωρισμένε ενώσει και θα έπρεπε και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να υπάρχει ένα κώδικα διοντολογία για τα πολιτικά κόμματα και να μην λησμονούμε και τα συνδικάτα. Διότι όσον αφορά το τι το δεν γνωρίζει κανεί τι γίνεται τι, στι χώρε μα, ε, στη χώρα μου τουλάχιστον έχουν το παγκόσμιο ρεκόρ. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο. Μια διευκρίνηση στα όσα είπατε κι εσείς για τη χρήση των κονδυλίων από πλευράς ε, οργανωμένου εγκλήματος. Προχθές είχαμε μια επιχείρηση της, ε, τους ΔΟΕ στην ε, Σικελία Από το 2004 στο 2009 χρησιμοποιήθηκαν 230.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια από τον ε, επικεφαλής ε, της μαφίας ε, στη Σικελία, τον Σπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ουσιαστικά αυτά τα κονδύλια και θα πρέπει να βρούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν. Η κυρία Ιώτοβα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο δεν είναι εύκολο να προετοιμάσει κανείς μια τέτοια έκθεση μετά από τις διάφορες ακροάσεις ε, που είχαμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε ως αποτέλεσμα των ε, συναντήσεών μας ε, στην Ιταλία περιέχονται αλλά έχω εγώ να κάνω μια ερώτηση και κάποια συμπεράσματα να βγάλω πρώτα απ' όλα ο κ. Γιακολίνου θα έπρεπε ίσως να ξεκαθαρίσει γιατί έχει συμπεριλάβει στον ορισμό της διαφθοράς την έννοια της πρόθεσης ή υπόσχεσης διαφθοράς. Στέκει αυτό το πράγμα στο δικαστήριο. Δεύτερον, υπάρχει κάτι το οποίο λείπει και αποτελεί μια σημαντική πηγή διαφθοράς ε, νομίζω. Τρίτον, η έκθεση αναφέρει ειδικού κώδικες ε, πολιτικών κομμάτων, επιχειρήσεων κτλ. Έχουμε από τη Βουλγαρία. Έχουμε τέτοιους κώδικες, αλλά μόνο στα χαρτιά. Και σπανίως έχουν ε, κάποιο αποτέλεσμα ή τους λαμβάνει ο κόσμος υπόψη. Νομίζω πως ε, θα πρέπει οι συστάσεις να είναι πολύ πιο κατηγορηματικές από έναν κώδικα συμπεριφοράς. Και τέλος το θέμα της πολιτικής ε, διαφθοράς. Πιθανώς δεν επαρκεί η διεφθαρμένη πολιτική να μην μπορούν να ξανακαταλάβουν ε, δημόσιες θέσεις. Ε, συχνά οι δικαστικές υποθέσεις ε, είναι μακροχρόνιες, ε, επέρχεται και παραγραφή και αποτελέσματα έχουμε πολύ σπάνια. Και υπάρχει κάτι πολύ ενισχυτικό όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς θα κόψουμε το γόρδιο δεσμό εάν χρησιμοποιούν τα κόμματα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, για να χρηματοδοτήσουν την πολιτική τους εκστρατεία, για να διαφημίζουν τα έργα που υποτίθεται ότι κάνουν και κατ' ουσίαν ε, πληρώνουν και δορδοκούν μίμιε και ανθρώπους. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πιο λεπτομέρως. Και θα πρέπει να υιοθετήσουμε μέτρα, κοινά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι κυβερνήσει των κρατών μελών να λάβουν υπόψη ε, τι ε, θέσει αυτέ και να μην εξακολουθήσουν οι πρακτικέ. Ευχαριστώ κυρία Ιώτοβα. Κύριε Γιακολίνο, έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφου που μου έδωσαν τη δυνατότητα να απαντήσω σε κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να εξετάσουμε λίγο περισσότερο στη διάρκεια της εισαγωγικής μου παρέμβασης. Να πω στον κύριο Νιούτον Ντάν ότι είναι σαφές ότι το θέμα αφορά την κορυφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κορυφή είναι σημαντική, αλλά παραδείγματο χάρη σε μια δημόσια διοίκηση όπου η τελική πράξη έχει προκύψει από μια βαθμιδών ε, ε, διαδικασία ε, μέχρι να φτάσουμε στην ευθύνη του επικεφαλής ίσως πρέπει να δούμε και τι έχει γίνει στην αρχή και το αντίθετο μπορεί ο πρόεδρος Σούλτ, όπως ανέφερε εσύ το παράδειγμά σου, αν είναι αυτό υπεύθυνο, θα έπρεπε να έχουμε και εμείς. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει τις οποίε το πρόβλημα δεν αφορά ε, των επικεφαλής. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, σίγουρα πρέπει να είναι αυστηρός ο έλεγχος, όπως έλεγε και ο κύριος Μποργέτσιο, πρέπει ε, να μας ενδιαφέρει όλο ένα και περισσότερο το θέμα της πρόληψης, αλλά εγώ θεωρώ ότι όλες οι διαδικασίες, για να αναφερθώ σε αυτό που ανέφερε και η κυρία Ιώτοβα, το τι γίνεται για την ε, κατανομή των πόρων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι πολύ καλές και να υπάρχουν και πάλι απάτη ε, και ε, να υπάρχει και ένα ενδιάμεσο στάδιο, αν θέλετε, ευθύνη σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και από την άλλη μεριά από αυτόν ο οποίος έχει σύμβαση με τη δημόσια διοίκηση. Τώρα, ορισμός της διαφθοράς. Εμείς κάναμε μια απόπειρα να ε, καταλήξουμε σε ένα ορισμό και ελπίζω, όπως ε, αυτό που είπε η κυρία Ιώτοβα, να είναι σαφή ε, και να αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά τους ορισμούς πρέπει να τους αξιολογήσουμε και πάντα φυσικά μπορούμε να τους βελτιώσουμε. Όσον αφορά τώρα αυτούς τους ε, αζάν προβοκατέρ, το θέμα της ευθύνης ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι παρόντες ε, σε ε, εγκλήματα τα οποία ε, ταράσουν την ε, κοινωνία, όπως για παράδειγμα το οργανωμένο έγκλημα. Και πρέπει να προβλέπεται και αυτή η δυνατότητα σε περίπτωση διεθνούς διαφθοράς, όταν συμμετέχουν περισσότερα κράτη-μέλη και θα μπορούσε να αποτελέσει και σημείο αναφοράς εάν το συνδέσουμε και με την δυνατότητα μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα ασχοληθεί και με τα θέματα αυτά και θα έχει δυνατότητες ανάκρισης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το έγκριμα, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να έχει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και οι τρεις συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο, ο κ. Μποργκέτσιο, ο Μπίλ και η κυρία Ιώτοβα, αναφέρθηκαν στο θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς, εύκολες διαδικασίες ε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουν πολλά κράτη-μέλη και σίγουρα θα περιλαμβάνεται και στην ενδιάμεση έκθεση. Τα έγγραφά μας, και εδώ αναφέρομαι τώρα στα έγγραφα όλης της Επιτροπής, ε, είναι ανοιχτά. Δηλαδή, πάντα δεχόμαστε βελτιώσεις και με την ε, σημαντική συνεισφορά των συναδέλφων και εγώ είχα πολύ θετικές συνεισφορές ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Σέβομαι πάντα τη Μεγάλη Βρετανία, Μπιλ. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα μοντέλο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν σε μια χώρα και πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, υπήρχε η εκλική εμπειρία που παρουσιάστηκε για την, ε, την παράθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πώς αντιμετώπισε την απάτη και το αναφέρω και αυτά κάπως στο έγγραφό μου. Και στην ε, Ηνωμένο Βασίλειο όμως και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες απαιτείται να βρούμε ένα μοντέλο κοινή επίθεση ε, απέναντι στα φαινόμενα τη διαφθορά και από εκεί και πέρα σε κάθε κράτο μέλο θα προσαρμοστεί ανάλογα με τι ιδιαιτερότητε και τι απαιτήσει τη κάθε χώρα. Για την υπόθεση Μπερλουσκόνη την έχουμε συζητήσει επανειλημμένω. Ο Μπίλ τον έχει ρωτευτεί, τον Μπερλουσκόνη. Και τον του ζητάτε να αναλάβει τι ευθύνε του. Στην Ιταλία υπάρχει η αρχή του ότι ο καθή θεωρείται αθώο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο στο Σύνταγμα που ε, ουσιαστικά θέτει τον Μπερλουσκόνη ισότιμο με τα υπόλοιπα 60 εκατομμύρια των Ιταλών. Ο κύριος Μποργέτσιο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εδώ βρισκόμαστε σήμερα για μια πρώτη προσέγγιση στη διαφθορά. Σίγουρα αποτελεί καλή εφαλτήριο, αλλά σίγουρα χρήση βελτιώσεων και η δική σας συνεισφορά σίγουρα θα βελτιώσει τα πράγματα. Όσον αφορά τη δυνατότητα να μην ξαναθέτει υποψηφιότητα κάποιο διεφθαρμένος πολιτικός, όλοι συμφωνούμε. Και η κυρία Αλφάνο άλλωστε είναι ε, άλλωστε γνώστης του θέματος και θεωρεί ότι όπως θεωρώ και εγώ ότι όποιος έσφαλε πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα κατάλογο Σήμερα χρησιμοποιείται και ο όρος που το ξέρει και ο κύριος ε, Ταταρέλα, έφυγε βέβαια, ήταν εδώ, ε, ατόμων που είναι ακατάλληλοι, δεν πρέπει να παρουσιάζονται σε εκλογέ. Ή θα πρέπει λοιπόν να για μία θητεία να μην μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ή να πρέπει να παραμείνουν εκτός εκλογικής διαδικασίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κατά πόσο θα είναι μόνιμη αυτή η να πρεπει να παραμεινουν εκτος εκλογικη διαδικασια τωρα ή προσωρινή θα το αποφασίσει η Επιτροπή, τα αφήνω σε εσά. Ευχαριστώ, διότι απαντήσατε και στις ε, ε, ε, σκέψεις μου και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την παρέμβασή τους. Ε, κύριε Αλφάνο, ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το πρώτο στάδιο της ανταλλαγής απόψεων. Ο κύριος Νιούτον Τάν αναφερόταν στις ε, οριστικές καταδίκες ε, που ε, υπάρχουν για την υπόθεση Μπερλουσκόνη. Είναι σαφές ότι υπάρχει η αρχή της αθότητες, αλλά υπάρχουν διάφορες οριστικές τελεσίδικες αποφάσεις και αυτές θα πρέπει να, να δούμε. Υπάρχει ένας δικαστής τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ η Ιταλία και τον σκότωσε η μαφία και ο οποίος έλεγε ότι πριν από την τελεσίδικη απόφαση ενός δικαστηρίου υπάρχει και ηθική καταδίκη και σε εμά πολιτικούς λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει και ηθική κρίση και θα πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Ιακολίνο. Να περάσουμε τώρα στην ακρόαση ποινικό δίκαιο, ε, έρευνες ε, και ε, θέματα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Στο πρώτο ερώτημα στο πρώτο πάνελ είναι κατά πόσον χρειαζόμαστε μια πολιτική κατά της μαφίας στην Ιταλία. Θα ακούσουμε τον κύριο Στέφανο Μαρσερβίζη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα μας μιλήσει για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να νομοθετήσει ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Κατόπιν, μετά από την έκθεσή σου, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπιγκό, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Παρίσι και καθηγητής μελετών στο King's College του Λονδίνου και θα μας μιλήσει για το οργανωμένο έγκλημα ως πρόκληση για το ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15 λεπτά για τον καθένα. Να δώσω αμέσως το λόγο στο Γενικό Διευθυντή ε, Στέφανο Μασερβίση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, καλή χρονιά και σε εσά και σε όλη την Επιτροπή ΚΡΙΜ, η οποία κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά για να γίνω πιο εύκολα κατανοητός. Νομίζω πως ε, το θέμα το οποίο συζητάτε σήμερα έχει μεγάλη σημασία αφ' αυτό αλλά και στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η αυξανόμενη ολοκλήρωση σε οικονομικούς ε, όρους και διάφοροι παράγοντες ε, που υποτίθεται πώς ενισχύουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, στηρίζουν πιο πολύ την οικονομική και την πολιτική διάσταση. Ε, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίο γίνεται η συζήτηση. Άρα το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος ε, αφορά και ένα πεδίο το οποίο δεν είναι μόνο αυτό της εγκληματικότητας αλλά και την απειλή που αποτελεί η εγκληματικότητα για όλες τις προσπάθειες των πολιτών, των κρατών, των δημοκρατικών θεσμών για να αλλάξουν, να μετασχηματιστούν όπως θέλετε πείτε το. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για μια αυστηρά ε, εγκληματική διάσταση αλλά και για μια οικονομική διάσταση. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε με κάποιον ρεαλισμό αλλά και σκεπτόμενοι το μέλλον. Γιατί σχετίζεται με το τι γίνεται από την Ευρώπη και αλλού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Το 2011 παρουσίασε μια έκθεση που τόνιζε την ε, σημαντική απειλή που αποτελούν ε, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες από την πλευρά της Κομισιόν. Συμφωνούμε πλήρως με την ανάλυση αυτή και τονίζουμε κάτι το σημαντικό, ότι δηλαδή για εμάς το οργανωμένο έγκλημα είναι διεθνές. Όσο περισσότερο προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τόσο περισσότερο το εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα για να βγάλει κέρδη και να εξασθενήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Οπότε όταν λέμε πως ε, το οργανωμένο έγκλημα κίνηγα το οικονομικό όφελος, αυτό είναι μία μόνο πτυχή της πραγματικότητας. Ξέρετε πως ε, το οργανωμένο έγκλημα και η μαφία εξασθενίζει τις δημοκρατικούς ε, θεσμούς. Οπότε αμέσως ή εμέσως υπάρχει μία πολιτική διάσταση του οργανωμένου έγκληματος στο πλαίσιο αυτό που είναι η... ποια είναι η κατάσταση τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, συμπεριλαμβάνει και το οργανωμένο έγκλημα στο άρθρο 83.1 Οπότε έχουμε ξεκάθαρα μια νομική βάση για να δράσουμε. Και εδώ πέρα βέβαια έχουμε μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, γιατί αυτά τα οποία υπήρχαν αφορούσαν την κατάσταση ε, προ Λισαβόνας. Και άρα υπάρχει ένα κενό το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να καλυφθεί. Οπότε σε αξιολογήσουμε το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η Ένωση εδώ και χρόνια έχει υιοθετήσει νομοθεσία που ποινικοποιεί τη συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται για την απόφαση 2008-841 ε, η οποία καθιστά τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη-μέλη και ορίζει ελάχιστες ποινές. Γνωρίζετε την απόφαση πλαίσιο, δεν θα την περιγράψω. Θα ήθελα να αναφέρω τα βασικά σημεία κριτικής. από και πανεπιστημίων αλλά και ανθρώπων που ασχολούνται σε καθημερινή βάση με το θέμα. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση αυτή δεν αρμονίζει πλήρως την έννοια της εγκληματική οργάνωσης και των εγκληματικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται. Οπότε, ε, ξέρετε, υπάρχουν κάποια όρια. Έχει μία ένα πολύ περιορισμένο ορισμό και άρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι χρήσιμη. Κατά την άποψή μας γνωρίζετε πως η άποψη αυτή πλαίσιο υιοθετήθηκε σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Υπήρχαν κάποιες φιλοδοξίες της Κομισιόν, οι οποίες βέβαια στη διαδικασία από το Συμβούλιο μετριάστηκαν. Και τότε η Ιταλία μας με κάποιες άλλες χώρες ε, έκαναν μια δήλωση λέγοντας πως το αποτέλεσμα ήταν ε, μέτριο. Οπότε, τι κάνουμε από εδώ και προς. Πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνουμε πως καλύπτονται οι εγκληματικές οργανώσεις ε, με σταθερή οργάνωση και δομή. Και δεν είναι απλά συνεργή σε ένα έγκλημα. Επιπλέον τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και άρα Ε, και τα κράτη-μέλη εδώ πέρα μπορούν να κάνουν ε, ό,τι θέλουν. Είναι το, με ένα σύστημα κάπως à la κάτι το οποίο βέβαια ίσχυε πριν από τη θέση της συνθήκης αγώνας. Και τέλος υπάρχει το κατόφλι των τεσσάρων ετών ε, φυλάξης που είναι ένα όριο. Η κριτική λοιπόν που ασκείται εδώ πέρα είναι σωστή. Εμείς συμφωνούμε. Το είχαμε πει βεβαίως και με την ε, δήλωσή μας. Όχι μόνο ε, γιατί οι προτάσεις μας ε, κάπως εξασθένησαν, αλλά αν δείτε και την σύμβαση του Παλέρμο έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. υπάρχει δηλαδή μια ζώνη ελευθερίας και ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Όπως προβλέπετε στην απόφαση, προετοιμάζουμε μία έκθεση για να δούμε ανεξαρτήτως του περιεχομένου την κατάσταση όσον αφορά την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Η έκθεση αυτή θα εγκριθεί αργότερα εντός του έτους και θα είναι αντικειμενική, θα εκθέτει τα γεγονότα όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και τις αδυναμίες. Γιατί, πέρα από αυτά τα στοιχεία, πολλά κράτη-μέλη πέσαν πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές. Οπότε είναι κάπως κακή η κατάσταση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, όπως ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινήσαμε και μία σχετική μελέτη και για τις ειδικέ ερευνητικέ πρακτικές και για το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος και με βάση αυτές τις δύο μελέτες και πιθανώς το, τη δουλειά της Επιτροπής σας θα δούμε το τι θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Βεβαίως, στο ενδιάμεσο δεν σταματήσαμε τις δραστηριότητες μας γιατί είχε αλλάξει η νομική βάση και βασιζόμενη στην συνθήκη της Λισαβόνας προτείνουμε τώρα κάποια άλλα μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν διαφορετικές πτυχές. Γνωρίζετε την οδηγία για την δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Αναγνωρίζουμε πως είναι μία μερική προσέγγιση, αλλά στοχεύουμε στα κέρδη της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Χτυπάμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Δυστυχώ, οφείλω να πω πως και εδώ πέρα το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με αυτό το οποίο είδαμε στην απόψη πλαίσιο το 2008. Γιατί διαρκώς οι συζητήσεις είναι ε, όλο και λιγότερο φιλόδοξες. Θα υπενθυμίσω εδώ πέρα την τεράστια συζήτηση για την ε, Επιτροπή ε, ε, που αντικατοπτρίζει όλες τις εμπειρίες των κρατών μελών και έχοντας ακούσει και όλες τις ε, υπηρεσίες ε, δίωξης. Ναι, είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά δεν πρέπει και να αποκλίνουμε από τον πραγματικό μας στόχο. Οπότε το προτείναμε αυτό, προτείναμε αυτή την προσέγγιση, η οποία είναι συνολική, γιατί ε, πρέπει, όπως είπα, να χτυπήσουμε, πρέπει να χτυπήσουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά σας προειδοποιώ πως δεν πάμε ακριβώς στην επιθυμητή κατεύθυνση. Δεύτερον, μια άλλη πρόταση. Έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογή για το αδίκημα του να πλήττει κανείς τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας. Κατόπιν έχουμε το ξέπλυμα χρήματος, όπου θα υπάρξει μια περαιτέρω εναρμόνιση του ορισμού και τρίτον να αναφέρω και την πρωτοβουλία μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε και το ξέρετε καλύτερα από μένα είναι πως ε, το οργανωμένο έγκλημα και ειδικά οι μαφιόζικες ομάδες δεν είναι μόνο μονοδιάστατες, δεν είναι μόνο μια ομάδα η οποία ληστεύει μια τράπεζα ή επιτίθεται σε μια τράπεζα. Είναι μια ομάδα η οποία διεισδύει στην οικονομία, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και έγκλημα με τη στενή έννοια. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Για το μέλλον, τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα ας προσπαθήσουμε να βγάλουμε ό,τι μπορούμε από την διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Έχουμε αρκετά υψηλές φιλοδοξίες για την οδηγία δίμευσης, ε, για την ανάλυση την τρέχουσα, για το τι γίνεται με το ξέπλυμα του χρήματος, αλλά νομίζω πως υπάρχουν στοιχεία για να καταδείξουμε πως, όπως είπα στην αρχή, όσο πιο πολύ προχωράει η ολοκλήρωση και παλεύουμε με την ανεργία και τις κοινωνικές ανταρχές, τόσο πιο πολύ ευνοείται το οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερον, όλοι ξέρουν ή θα έπρεπε να ξέρουν πως οι μαφίες δεν είναι τοπικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό. Δείτε τι γίνεται σε μια χώρα όπως η Ιταλία, ε, που συχνά θεωρείται το κέντρο βαρύτητας της μαφίας. Ε, η μαφία δεν είναι νότιο ζήτημα, υπάρχει και στο βορρά, σε όλα τα κράτη-μέλη. οπότε είναι κοινό πρόβλημα. Εάν δεν έχουμε κοινή νομοθεσία, κοινέ προδιαγραφέ, δεν θα το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Το δεύτερο λοιπόν είναι αυτό, δεν είναι τοπικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο και οπωσδήποτε ευρωπαϊκό. Μετά το προσεγγίζουμε τομέα. Τομέα προσπαθώντας να βρούμε τις διαφορετικές πτυχές. Αυτό είναι σημαντικό και βεβαίω έχουμε υποχρέωση να έχουμε αποτελέσματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι αποτελεσματικό. Και υπάρχει, θα έλεγα, ένα μεγάλο κενό, μια απόκληση μεταξύ της πολιτικής συζήτησης και της πραγματικότητας όταν φτάνουμε σε συγκεκριμένα νομοθετήματα. Γιατί δεν υπάρχει συνέχεια με το τι διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή περιδίμευσης και της ε, ενημέρωσης στο υψηλό πολιτικό επίπεδο. Γιατί συνεχώς μειώνονται οι φιλοδοξίες. Πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Εγώ προτείνω να κοιτάξουμε μια κατεύθυνση. Ξέρετε, είναι προφανές ότι από τώρα μέχρι το τέλος της ε, θητείας ε, και την εφαρμογή του προγράμματος Στοκχόλμης έχουμε, έχουμε πολύ ε, περιορισμένο πλαίσιο αλλά προτείνω ειδικά στην Επιτροπή σας να κοιτάξει να δει το τι μπορεί να γίνει μετά τη Στοκχόλμη κάτι το οποίο δηλαδή θα ξεκινήσει το 2015 αν τηρήσουμε όλες τις ε, προθεσμίες και νομίζω πως ε, αυτό θα ισχύσει για να δούμε έτσι με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο αυτά τα φαινόμενα και να πούμε πως εφόσον σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα δώσει κάποιες κατευθύνσεις εάν στα έγγραφα αυτά η πτυχή αυτή της ε, πολλαπλότητας ε, του οργανωμένου εγκλήματος και του μαφιόζικου φαινομένου συνδυαστεί με την ανάγκη ε, παροχής προσθέμενης αξίας σε εθνικό επίπεδο, ίσως μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι πιο φιλόδοξο. Αυτές είναι κάποιες μικρές προτάσεις, καθώς τώρα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον. Ε, επιτελείται τώρα το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, οπότε το 2014 θα ξεκινήσει μια διαδικασία και θα πρέπει η Επιτροπή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, να κάνει κάποιες προτάσεις. Και εμείς ευχαρίστως βεβαίω να το δεχτούμε, θα καταθέσουμε κάποιες ιδέες. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να τα συζητάμε αυτά ε, για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την πολύ σημαντική κατεύθυνση. Ευχαριστούμε όχι μόνο για τη σαφήνειά σας και τη διαφάνεια στη διάρκεια της παρουσίασης, αλλά γιατί μας παρουσιάσατε τα διάφορα προβλήματα και μας προσφέρετε και κάποιες πιθανές λύσεις. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά την παρέμβασή σας. Οι σκέψεις σας είναι μοχλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εσείς ε, που λέτε και υποστηρίζετε ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι να έχει ενιαίους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους ε, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από νομική σκοπιά σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, ακριβώς και για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφάλειας ε, των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι διότι μας αφιερώσετε το χρόνο σας. Να δώσω τώρα το λόγο για 15 λεπτά στον καθηγητή Didier Μπίγκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω μια έρευνα δική μου αλλά και τριών ακόμη συνεργατών μεταξύ του οποίων ο καθηγητής Σέπτη και η κυρία Μπέντζαφερ έχει ήδη δημοσιευθεί και θα προσπαθήσω μόνο απλώς να σας παρουσιάσω τα κυριότερα σημεία που μπορεί να ενδιαφέρουν και εσάς. Ένα από τα σημαντικότερα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ανάλυση των εξελίξεων του ορισμού του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Έχουν ακουστεί με πολλές κοινοτοπίες ορισμοί τόσο μπανάλ που κανείς πια δεν αναρωτιέται τι παίζεται όταν μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα τι σημαίνει ακριβώς το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα μιλώντας βέβαια πάντο για σοβαρά εγκλήματα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας δείξω ότι η απλή επανάληψη του ορισμού του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος δεν λύνει το πρόβλημα που είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι λέμε συνήθως και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λάθος ανάλυση. Το δεύτερο τμήμα της ερευνάς μου αφορά τι είδους πολιτική και προσέγγιση μπορεί και πρέπει να αναλάβουμε ποιος θα είναι ο ρόλος μιας ειδικευμένης ενωσιακής αστυνομίας αλλά και της νομοθεσίας και ο ρόλος των τοπικών αρχών. Ποιες ανάγκες υπάρχουν ανατομέα ας πούμε. Βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι δεν είναι καινούριο πρόβλημα το οργανωμένο έγκλημα. Θα θυμάστε την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στα ΣΥΠΑ. Και αυτό το λέω γιατί ήδη από την αρχή ο ορισμός της δραστηριότητας των παρανόμων ομάδων που παρήγαγαν ενόπνευμα είχε τεθεί ως πρόβλημα. Στο τέλος της δεκαετίας του 70 υπήρξε μία διπλή εξέλιξη. Πρώτα, de facto μείωση της ε, παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και οι αναλυτές το διαχώρισαν από την διαφθορά λέγοντας ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, αφορά εγκληματίες που προέρχονται από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνίας ενώ ταυτόχρονα παρατηρούσαν ότι το οργανωμένο έγκλημα διευρύνεται και ότι πετυχαίνει επειδή είναι διαμεθοριακό και διεθνικό. Από το διεθνές λοιπόν οργανωμένο έγκλημα περάσαμε στην έννοια του διαμεθοριακού και υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Έννοια η οποία συνεχίστηκε να αναπαράγεται και από τις Ηνωμένε Πολιτείες και τη δεκαετία του 90. Μερικές χώρες έλεγαν ότι μέσα στην κοινωνία τους υπήρχαν τα στοιχεία αυτά και άλλες που δεν ήταν σίγουρες αν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η ορολογία που ανέφερε τη μαφία. Ίσως λοιπόν ένα από τα στοιχεία που πρέπει να αναφερθεί εδώ σύντομα είναι ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 και τα τέλη του ψυχρού πολέμου τι έγινε με το οργανωμένο έγκλημα. Μια αλλαγή. Όλο και λιγότεροι ανθρωπολόγοι και εγκληματολόγοι ασχολούνταν με αυτό και όλο και περισσότεροι που ανελάμβαναν στρατηγικές μελέτες ή μελέτες στρατηγικής, διότι το οργανωμένο έγκλημα το θεωρούσαν σαν θέμα στρατιωτικής περίπου στρατηγικής. Έλεγαν δηλαδή ότι οι εγκληματικές ομάδες μπορούν να αναλυθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι στρατιωτικές εισβολές. Αυτό έγινε της μόδας. Είδαμε πολλούς αναλυτές και άτλαντες γεωπολιτικούς του εγκλήματος. Να ένας εδώ. όπου προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι η επικίνδυνότητα του φαινομένου έγκυται στην καθολικότητά του. Ένας και μόνο χάρτης λοιπόν δίνει την εντύπωση ότι όλα είναι σφαιρικά και καθολικά. Έτσι όμως συνδυάζουμε υπερβολικά, ταυτίζουμε μάλλον, συγχαίουμε την εικόνα, πραγματική εικόνα του οργανωμένου κλίματος. Γιατί, γιατί διαστρεβλώνεται έτσι η πραγματικότητα. Το έγκλημα είναι στρατιωτική απειλή. Αυτό πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα. Έτσι θα το δούμε ή ως θέμα αστυνόμευσης και δίωξης ή γενικότερης οργάνωσης της κοινωνίας. Οι περισσότεροι τέτοιοι χάρτες συνέχεια ανεπισης ορισμένες εγκληματικές οργανώσεις με εθνοτικές οργανώσεις, ας πούμε το κινέζικο οργανωμένο έγκλημα, το αφρικανικό οργανωμένο έγκλημα. Τι σημαίνει όμως αυτό. Έτσι δημιουργούμε μια επικίνδυνη τάση κατά ορισμένων κοινοτήτων ολοκλήρων και όχι κατά των πραγματικών υπεύθυνων του εγκλήματος. και κρύβουμε το σημαντικότερο στοιχείο που είναι η τοπική διάσταση του εγκλήματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία πολύ ισχυρή τοπική διάσταση του οργανωμένου εγκλήματος και ότι κάθε περίπτωση πρέπει να αναλύεται μεμονωμένα. Φυσικά οι τοπικοί εγκληματικοί παράγοντες πετυχαίνουν γιατί γνωρίζουν την κοινωνία τους πολύ καλά. Αυτό είναι προφανές. Αλλά πολύ συχνά ξεχνιέται. Ξέρουν ποιες είναι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και αυτό τους δίνει ευκαιρίες. Όλο και περισσότερη έρευνα λοιπόν αναλήφθηκε ιδίως από τον Χόμπς και τον Πίτερ Ρόιτερ, που έλεγε ότι ναι υπάρχει μεν οργανωμένο έγκλημα αλλά υπάρχει και ανοργάνωτο έγκλημα το οποίο είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι εφήμερο αλλά πολύ σημαντικό. Και ο Βαρέσε επίσης στο βιβλίο του λέει ότι υπάρχουν μεν μαφίες αλλά δεν είναι και τόσο διεθνής γιατί υπάρχει ο γλωσσικός φραγμός. Υπάρχει, υπάρχουν τέτοιες μαφίες, αλλά δεν εξηγούν όλο το φαινόμενο. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Πρέπει να δούμε πολύ περισσότερο μορφές πολύ σοβαρού εγκλήματος που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην έννοια του μαφιόζικου τύπου οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι θα βλέπαμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες εγκληματικής δραστηριότητας που είναι εξίσου σημαντικές. Και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο ποιες είναι αυτές. Είναι η κοινωνική ζημία. Αν θέλουμε να συζητήσουμε τι είναι το σοβαρό έγκλημα, τότε πρέπει να μιλήσουμε για την κοινωνική ζημία που προξενεί γιατί έτσι μπορούμε να συζητήσουμε το, τα εγκλήματα αστικού τύπου, όχι μόνο από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνίας. Μπορεί να είναι λιγότερο βίαιες οι δραστηριότητες τους και άρα λιγότερο ορατές για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τους δημοσιογράφους, αλλά είναι πολύ σοβαρές περιπτώσεις αν εξετάσουμε το πόσο βλάπτουν το συμφέρον του πολίτη και της Ένωσης ολόκληρης. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους το έγκλημα. Μπορούμε να το δούμε συνοπτικά όπου διακρίνουμε τουλάχιστον τρία επίπεδα. Πρώτον της γενικής νομοθεσίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα ήταν εύκολο να ξέρ, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα αν ξέραμε εκ των προτέρων τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο γιατί δε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν μια τελείως νόμιμη επιχείρηση δρά παράνομα. Άρα η πρώτη δραστηριότητα που πρέπει να αναλάβουμε είναι η γενική νομοθεσία παραδείγματος χάρη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα ή η μετατροπή ορισμένων χρηματοπιστωτικών κέντρων σε φορολογικούς παραδείσους. Ίσως να είναι ακόμη πιο σημαντικό αυτό από ότι η ίδια η αστυνομική δουλειά. Το δεύτερο επίπεδο βέβαια είναι η αστυνομική δουλειά. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που ειδικεύονται στην καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου κλίματος και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις και υπηρεσίες. Αν όμως περιοριστούμε, αν όμως τους ζητήσουμε να τα κάνουν όλα από μόνοι τους δεν θα πετύχουν τίποτα. Άρα υπάρχει και το τρίτο επίπεδο, οι διοικητικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται την καθημερινή ζωή στις πόλεις. Τι διασύνδεση μπορούμε να δούμε μεταξύ αυτού του επίπεδου και του ευρωπαϊκού. Ας πούμε η Ευρωπόλ ήδη ασχολείται με ειδικευμένη αστυνομική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια αναδιοργάνωση του τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το επίπεδο της, την αναδιοργάνωση, για την αναδιοργάνωση της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα παράδειγμα θα ήταν ότι οι ειδικευμένες αστυνομικές μονάδες περιορίζονται στο να χειριστούν ορισμένα μόνο φαινόμενα και άρα δεν μπορούν να χειριστούν τα υπόλοιπα. Ίσως εδώ πρέπει να γίνει κάτι. Η γνώση της τοπικής κοινωνίας λοιπόν είναι απολύτως ζωτική. Τώρα, ποιες είναι οι δυσκολίες. Σίγουρα μέχρι πρόσφατα με την έκθεση Όκτα χειριστήκαμε μόνο μερικές ειδικευμένε ε, αστυνομικές υπηρεσίες που συνεννοούνταν μεταξύ τους. Τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή, ένα άνοιγμα και σε άλλους τομείς και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των ειδικών αλλά να μην είναι μόνον οι ειδικοί αυτοί εκείνοι που επιλέγονται από την Ευρωπόλ. Υπάρχουν λοιπόν εναλλακτικές λύσεις. Ας πούμε ο Σλέιπνιρ από τη Royal Canadian Mountain Police που τονίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων τύπων σοβαρού εγκλήματος και λέει ότι ένα από τα κριτήρια πρέπει οπωσδήποτε να είναι και η κοινωνική ζημία. Το... Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ένας ενωσιακός νόμος κατά της μαφίας, σοβαρό θα ήταν μεν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλη την ποικιλομορφία του φαινομένου και ο νόμος αυτός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο το συνήθι τύπο εγκλήματος αλλά και το κοινωνικό έγκλημα σε πλήρη συνεργασία με, την τοπική, με τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Μπηγό. Να ξεκινήσει η συζήτηση και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Ταβάρες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Παρουσιάσεις ε, γενικής ε, και ειδική φύσης και με πολύ καλές ιδέες ε, για το μέλλον. Και μια που είναι εδώ πέρα ο κύριος θέλω να τον ρωτήσω κάποια πράγματα που ήταν ε, ε, κομμάτι της δουλειά μας όταν συζητούσαμε την οδηγία δίμευση, δηλαδή το ζήτημα της καταδίκης ήμι και το θέμα του ορισμού της ε, του παγώματος ε, ή της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σαφώς υπάρχουν πολλές αμφιβολίες μεταξύ των συναδέλφων για το ότι θα μπορούσε θα μπορούσαν να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία κάποιου χωρίς καταδικαστική απόφαση και με βάση τον, ορισμό του τρόπου ζωής που ήταν μία από τις εκφράσεις που είδαμε εκεί πέρα βεβαίως ξέρουμε πως ο ορισμός αυτός ε, προέρχεται από την, ε, τον κοινωνιολογικό ορισμό της μαφίας αλλά βεβαίως υπάρχει τεράστια πιθανότητα κατάχρησης ε, Π.χ. μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτικές απόψεις και να τις θεωρήσουμε ως τρόπο ζωής. Οπότε, θα ήθελα εσείς ε, να μου απαντήσετε σε αυτό. Γιατί υπάρχουν αμφιβολίες, επιφυλακτικότητα και στο Συμβουλίο που οπωσδήποτε θα, θα εξασθενήσει την νομοθεσία ε, Καταλαβαίνω τις ανησυχίες της Κομισιόν, αλλά οπωσδήποτε δεν θα αντιμετωπιστούν έτσι οι σοβαρές ανησυχίες που έχουμε κι εμείς. Ίσως ένας σαφέστερος ορισμός ε, των διαφορών ε, παγώματος και κατάσχεσης ε, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Δηλαδή μπορεί να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων που δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά όχι να κατασχεθούν. Αλλιώ ανησυχώ πως δεν θα υπάρξει καμία συνένεση. Σε τι μπορούμε να έχουμε συνένεση τώρα. Στον τομέα το τραπεζικό. Και πολλά προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να γίνει πιο δύσκολο για τις εγκληματικές οργανώσεις να βάλουν σε τράπεζες τα περισσιακά του στοιχεία. Προφανώς δεν επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια οι τράπεζες και πρέπει να νομοθετήσουμε για να γίνει αυτό για να ξέρουμε ποιοι είναι οι τελικοί ιδιοκτήτες ε, δικαιούχοι, πώς θα το πείτε, ε, των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Και κάτι το οποίο θεωρώ πως η Κομισιόν θα πρέπει ε, στο πλαίσιο της σκέψης μας αυτής, στο πλαίσιο δηλαδή του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού να υπάρξει μια μονάδα διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είτε με την Europol, αλλά μετά υπάρχει και κάτι άλλο πρέπει να δούμε, δηλαδή τι σχέση θα έχει η Ευρωπόλ με το Κοινοβούλιο. Σαφώς δεν είναι ικανοποιητική η σχέση. Στη Λίμπε, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές ε, έρχονται άνθρωποι από τους, της Europol και δεν μας ε, δίνουν τις πληροφορίες. Και δεν είναι και υποχρεωμένοι από το νομοθεσία. Οπότε είναι ένα ζήτημα... Ε, αν συγκρίνει κανεί ας πούμε, το, το τι γίνεται με το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ε, δεν μπορεί κανεί να πάει και να αρνηθεί να καταθέσει ή να δώσει παραπλανητικέ πληροφορίε είναι έγκλημα. Okay. Εδώ πέρα έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μα δίνουν και παραπλανητικέ πληροφορίε. Okay. Οπότε, αν είναι να τους δώσουν περισσότερε ε, εξουσίε, χρειάζεται και περισσότερο έλεγχο. Ήθελα λοιπόν επίσης να αναφέρω και κάποια πράγματα για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση του καθηγητή του κυρίου Μπίγκο. Οπωσδήποτε ένα νόμο ο οποίο δεν έχει συνταχθεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ζουν χάρη τι έγινε με την ποταπαγόρευση στη ΣΥΠΑ. Εκεί πέρα δημιουργήθηκε περισσότερο έγκλημα. Οπότε ε, δημιουργείται έτσι και διαφθορά και διάβρωση της δημοκρατικής πολιτείας που είναι κάτι το σημαντικό και φοβάμαι πως ε, αυτό δημιουργούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη θυμήθηκα και το παλιό εβραϊκό αστείο με το γέρο που λέει «Καλωσορίζω την άφηξη του οργανωμένου εγκλήματος στο Ισραήλ γιατί είναι το πρώτο οργανωμένο πράγμα που βλέπω στη χώρα». Ε, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα μια πολιτεία η οποία βασίζεται στην, σε αρχές. Γιατί πάντα αντιδρούμε ως αστυνομικοί σε κάποιες απειλές, αντί να έχουμε κάποιες αρχές. Οπότε είναι σαφές αυτό το οποίο είπατε βέβαια για την κοινωνική ζημία. Αλλά σκέφτηκα κάτι τρομακτικό. Εάν ορίσουμε το οργανωμένο έγκλημα ως κοινωνική ζημία, μήπως τα θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις δεν είναι μέρος του. Έχω δει εγώ α, τα θεσμικά όργανα να προκαλούν την περισσότερη κοινωνική ζημία τα τελευταία χρόνια. Είναι λοιπόν οργανωμένο έγκλημα. Πώς το ορίζουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σε ένα τόσο ευρύ πλαίσιο το να εντοπίσουμε και στα πλαίσια της συζήτησης που κάνουμε και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την Οδηγία για τη Δήμευση Περιουσίας και είναι και ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και στη χώρα μου τις δικαστικές αρχές και υπάρχουν σχεδόν καθημερινές αντιπαραθέσεις. Θα ήθελα να πω λοιπόν δύο λόγια προς υπεράσπιση της Europol. Η Επιτροπή μας με τη Europol μέχρι σήμερα είχε εξαιρετικές ε, σχέσεις, είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή πληροφοριών και τον επόμενο μήνα θα πάμε και στη Europol και στη Eurojust ε, με αποστολή και πρέπει να σας πω ότι πήγα και σε μία άτυπη επίσκεψη που ήταν και προσωπικό κίνητρο αλλά και πρόσκληση στη Washington στην οποία συμμετείχε και η Europol και ε, πρέπει να πω ότι όταν πήγαμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στη Washington ε, μιλήσαμε και για τη μελλοντική επίσκεψη που θα κάνουμε στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου στη Washington. Νομίζω ότι υπάρχουν οι καλές προθέσεις σίγουρα για μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά για το θέμα αυτό και ελπίζω τα προβλήματα τα οποία ανέφερε σε Σύρουη για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών με τη Europol να επιληθούν, διότι ε, η Επιτροπή πολιτιστικών Ελευθεριών είναι η μητέρα της Επιτροπής ΚΡΙΜ και θα πρέπει ε, να πούμε ότι τα προβλήματα με τη Europol δεν αφορούν εμάς. Εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους και όχι μόνο ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αλλά μπορώ να σου πω ότι την περασμένη εβδομάδα πήγα στην Νάπολη Ξέρετε, συνάδελφοι, ότι έγιναν σημαντικές επιχειρήσεις ε, καταπολέμησης της μαφίας από την ε, ανακριτική μονάδα καταπολέμησης της μαφίας και από την ε, εισαγγελία καταπολέμησης της μαφίας της Νάπολης. Il ruolo, ancora una volta, Και προκύπτει για άλλη μια φορά το εξή. Εμείς προσπαθούμε να συνδέσουμε Όλου του οργανισμούς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Από πλευράς τους υπάρχει σχετικό αίτημα να μπορέσουν να έχουν μία επικοινωνία. Πολύ συχνά ε, περιοριζόμαστε απλώ στην ανταλλαγή καλών πρακτικών. Πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα. Διότι πέρα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών πρέπει να υπάρχει μια ροή πληροφοριών, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για τη ροή των πληροφοριών και αυτό το οποίο προκύπτει από τις συναντήσεις που κάνω εγώ αυτούς τους μήνες, από τότε που έχω αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής ΚΡΙΜ, είναι ε, πάντα το εξή. Είναι πάντα όλοι οι οργανισμοί εκεί, η Europol, η Eurojust, ε, η ODC, αλλά ορισμένες φορές δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, κάποιες ε, φορές κάποιες πληροφορίες δεν διαβιβάζονται εντός ε, των ε, οργανισμών αυτών και δεν διαβάζονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι που ο Διευθυντής Μαρσερβιζή μας είπε ότι αυτή η Επιτροπή θεωρείται ως μια Επιτροπή που όχι μόνο πρέπει να παρουσιάσει ένα κείμενο, αλλά ως κάτι το οποίο μπορεί να ενώσει, όχι μόνο να συντονίσει, αλλά να διευκολύνει ε, ροή πληροφοριών και μια συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ όλων αυτών των οργάνων. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, ε, ιδίω όταν το αναγνωρίζουν άλλοι. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ιακολίνη. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μανσερβίζε. Πολύ ευθεία ερώτηση. Έχει προχωρήσει ιδιαίτερα το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και από ό,τι λέγεται μέχρι την Άνοιξη θα πρέπει να έχουμε έτοιμο το νομικό έγγραφο και να ε, υποβληθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ποια θα είναι η σχέση μαζί τους και για ποια δικήματα θα είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχετε στην παρούσα φάση ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μπιλ Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ναι. και είναι κρίμα το ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο mm. να τις δούμε και πιο λεπτομερώς. Ο κύριος ε, Μαντσεβίση, τον έχει ξανακούσει και θέλω να τον ξανακούσω είπε σωστά πως ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι πως οι Υπουργοί και το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο κάνουν το ελάχιστο. Τα νερώνουν, μιλάνε και κάνουν το απολύτως ελάχιστο. Αυτό δεν επαρκεί γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να βρούμε είναι ένας τρόπος να τους πιέσουμε να δράσουν. Και αυτό θα γίνει με το να κινητοποιήσουμε το κοινό και το κοινό θα πει στους ηγέτες σταματήστε να κάθεστε στις πολυθρόνες και κάνετε κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπει ο κόσμος και τηλεόραση και ταινίες ε, και τα λοιπά. Το να ενημερώσουμε το κοινό. Ε, είχα πριν από λίγα χρόνια μια συνομιλία με τον πρώτο διευθυντή της Europol ε, που λέει ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, πώς θα κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Και λέει ίσως χρειάζεται μια 11 Σεπτεμβρίου. Ε, λέει δεν το θέλω κάτι τέτοιο. Ε, οπότε δεν είναι λύση αυτό. Οπότε μια λύση που έχω να προτείνω για να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη είναι εάν η Κομισιόν έχει να προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού FBI. Θα είναι τόσο φοβερή αυτή η πρόταση. Θα αρχίσουν να ορλιάζουν τα ΜΜΕ, τα κράτη-μέλη και να λένε δεν γίνονται αυτά, αλλά θα ξεκινήσει μια συζήτηση και θα πει ο κόσμος γιατί και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα πούμε είναι διασυνοριακό το έγκλημα, δεν μπορούν να το παλέψουν οι αστυνομίε. Οπότε α κάνουμε μια δραματική πρόταση και αυτό είναι ο ρόλος της Κομισιόν. Εντάξει καλά, ε, θα σα πυροβολήσουν, αλλά δεν πειράζει, του χρόνου θα έρθει άλλη Κομισιόν και εσεί θα έχετε ακόμα τη δουλειά σα ελπίζω. Οπότε α προτείνουμε ε, ένα ευρωπαϊκό FBI να ξεκινήσει η συζήτηση και άρα ο ε, Ευρωπαϊκό. αυτό σημαίνει βεβαίως Ευρωπαϊκό Ποινικό Κώδικα Οπότε πείτε στον Επίτροπό σας να προτείνει ομοσπονδιακά μέτρα να ξεκινήσουμε. Ακόμα και αν δεν επιτύχουμε τίποτα στο τέλος, να ξεκινήσουμε τουλάχιστον. Και ε, κύριε καθηγητά, συναρπαστική η παρουσίασή σας και σας ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσετε να την στείλετε και στην Επιτροπή για να την διαβάσουμε. Αλλά ε, ε, βλέπω πως είστε καθηγητής... σε θέματα αμήνης ε, στο Λονδίνο. Ίσως μπορώ να έρθω στο Λονδίνο να τα πούμε κάποια στιγμή. Ε, θα τα πούμε. Ωραία, βλέπω ότι συγκατανεύετε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ναι, η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα στον κύριο Μανσερβίση. Εμείς ε, βεβαίως αναμένουμε την πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη διαφθορά εντός του έτους. Αν μπορούσατε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα, ποια θα είναι η δομή αυτής της έκθεσης. Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. και πώς συνεισφέρει στον κοινό μας στόχο για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο διεθνές επίπεδο. Και η δεύτερη μου ερώτηση, ο κύριο Μπίγκο. Συχνά συζητάμε για το πώς μπορεί να μετρηθεί το επίπεδο διαφθορά στα κράτη-μέλη. Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση η οποία όμως απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έλεγε πως δεν ήταν ε, αρκετά λεπτομερής η πρόταση, δεν είχε αντικειμενικά κριτήρια. Κρίνοντας ε, εσείς από την εμπειρία σας, ε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μετρήσουμε τη διαφθορά. Και τώρα ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ των όσων λέει ο συνάδελφος, ο Μπιλ, για το FBI. Ναι, εκπλήσεων που η Κομισιόν δεν κάνει περισσότερα. Γιατί, εάν δείτε τις έρευνες, τα ευρωβαρόμετρα κτλ. Βλέπετε πως υπάρχει στήριξη της κοινή γνώμης για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα ή το οποιοδήποτε έγκλημα. Και θα μπορούσατε ίσως να κάνετε μία μελέτη, να συγκρίνετε το τι συμβαίνει στην Αμερική και τι συμβαίνει στην Ευρώπη και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα οπωσδήποτε στη ΣΥΠΑ, αλλά τουλάχιστον εάν συγκρίνεται το μέγεθος, τη στελέχωση και τη δυναμικότητα, θα εκπλαγείτε. Σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι παρανυχίδα. Είναι και δική μας ευθύνη, όχι μόνο της Κομισιόν. Ε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Βεβαίω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ε, εγώ προέρχομαι από βόρεια χώρα, πώ έχουμε διαφορετικού πολιτισμού ε, στην Ευρώπη και αυτό είναι και κάποια προσθέμενη αξία. Σε άλλου τομεί βεβαίω δεν είναι. Γιατί κοιτάμε διαφορετικά το έγκλημα και βεβαίω αυτό είναι επίση μέρο του προβλήματο, αλλά αν ξεκινήσουμε με κοινούς ε, θεσμούς. Νομίζω πως έτσι θα καταπολεμήσουμε τα πιο σοβαρά προβλήματα. Ή τέλος πάντων οτιδήποτε συνέβη κατά τη διάρκεια των χαμένων ε, δεκαετιών. Για τον κύριο Μπίγκο. Ε, εξαπλάγει από τους ορισμούς οργανωμένου και ανοργάνωτου εγκλήματος. Νομίζω ότι και το οργανωμένο έγκλημα είναι κάπως ανοργάνωτο και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν κατάλαβα τα συμπεράσματά σας. Γιατί μιλάμε για οργανωμένο και ανοργάνωτο έγκλημα. Γι' αυτό αν είναι να μιλήσουμε για νομοθεσία, παραδείγματος χάρη για τα εγκλήματα μίσους, ε, συμφωνώ, αλλά αυτός ο ορισμός μετά έχει προβλήματα. Και ε, προς τον πρόεδρο, η αστυνομία παραδείγματος χάρη θεωρείται πως πρέπει να έρχεται εδώ πέρα και να αποκαλύπτει τα πάντα. Βεβαίω όχι να μας δίνει παραπλανητικές πληροφορίες, αλλά οι αστυνομίε. Ε, πρέπει να έχουν και κάποια μυστικά. Και να εργάζονται με τρόπο ανοιχτό. Ε, να μην παραπλανούν βεβαίω, Πρέπει να υπάρχει έλεγχο, Αλλά καμιά φορά είμαστε αφελεί. Και λέμε πώ πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Καμιά φορά. Και το κοινοβούλιο αυτό είναι σουρωτήριο όπω ξέρετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω αμέσω σε αυτό γιατί με ρωτήσατε εμένα. Ε, δεν λέω βεβαίω να αποκαλύψει κανεί λεπτομέρειε ε, ανοιχτών ερευνών. Αλλά γενικές πληροφορίες ε, σε αιτήσια βάση και ποιοτικές και ποσοτικές για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε καλύτερα και να επιβλέπουμε την εφαρμογή κάποιων διεθνών συμφωνιών που εμείς έχουμε θεσπίσει, νομίζω μπορεί να γίνει. Δεν θα αναπτύξω τώρα περαιτέρω. Σκεφτούμε παραδείγματος χάρη την εφαρμογή των συμφωνιών SWIFT που ψηφίσαμε και πρέπει να ξέρουμε περισσότερα για αυτές. Και γιατί δεν είχαμε ικανοποιητικές πληροφορίες για την πρόοδό τους. Και θα μείνω σε αυτά γιατί τα περισσότερα από αυτά τα οποία συζητάμε για αυτό το θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών και πρέπει να είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα έχουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών για να ξέρουμε σε τι έχουμε δεσμευτεί. Αυτό εννοώ. Η άποψή μου λοιπόν είναι πως η εντολή της Ευρωπόλ πρέπει να προσαρμοστεί για να υπάρχει περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος. Μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό, μια μέση λύση μεταξύ του να μην εμποδίζουμε τη δουλειά της αστυνομία, αλλά να ξέρουμε και αυτά που πρέπει να ξέρουμε ως εκπρόσωποι και νομοθέτες. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Εγώ τώρα πρέπει να φύγω, η Σόνια θα αναλάβει την Προεδρία, θα δώσει το λόγο στους καλεσμένους μας, αλλά σημειώνουμε οπωσδήποτε τις απαντήσεις σας, ειδικά για το ζήτημα της ε, δέσμευσης ή ε, κατάσχεσης ε, χωρίς καταδίκη. Μάλιστα. Θα δώσουμε ξανά τον λόγο στον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Μασερβίση για την απάντησή του. Ευχαριστώ. Καταρχάς, για το ζήτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Ταβάρες, για την... Ε, Όπω ξέρετε, η πρόταση της Κομισιόν για την εκτεταμένη κατάσχεση εφαρμόζεται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι περιορισμένη. Όταν εξετάζουμε τι προσπαθούμε να εναρμονίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο προβλέπει και εγγυήσει γιατί και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ίδια ασυμμετρία. Δεν πρέπει λοιπόν μόνο να έχουμε καλά ταυτισμένες περιπτώσεις, αλλά και να προβλέπουμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει επαρκέστερα η εναρμόνιση πανενοσιακός. Πάντα έτσι γίνεται. Ξέρετε ότι όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν καταχρήσεις, αλλά επίσης ότι αυτό είναι συμβατό με τις γενικές αρχές και την ομολογία όχι μόνο σε ενωσιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης που τα έχει αναλύσει και εκείνο αυτά και κατέληξε ακριβώς στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ορισμένες εγγυήσεις χωρίς εγγυήσεις ότι δεν θα παραβιαστούν δηλαδή τα ατομικά δικαιώματα. Τώρα, για την πιθανή αποσύνδεση μεταξύ ξεπαγώματος και αποκατάσχεσης. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και να δούμε και τι φρονεί σχετικώς η Ιρλανδική Προεδρία. Ίσως κάποιο συνδυασμό ποινικού και αστικού δικαίου για να καταλήξουμε στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Το στόχος είναι να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, η κυκλοφορία των χρημάτων, το κέρδος. Μπορεί να υπάρξουν διάφορα μέσα για να επιτευχθεί αυτό, αλλά να ξέρουμε τι ζητάμε. Μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορα εργαλεία, αλλά με τον όρο αυτός να είναι ο στόχος. Οι χώρες μέλη που έχουν νομοθεσία σχετικώς γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο. Ας υπάρξουν και εγγύησεις, αλλά να διατηρηθεί ο στόχος η κατάσχεση είναι επίσης σημαντική για να πάψει να παράγεται το κέρδος. Δεν μιλάμε μόνο για λεφτά, αλλά και για κτίρια, για οικονομικές δραστηριότητες, για κάτι που δεν είναι μόνο χρήματα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ναι, το πάγωμα χρημάτων είναι σημαντικό, αλλά χρειάζονται και τα υπόλοιπα. Πρέπει όλα αυτά να αποδοθούν και στην κοινωνία όχι μόνο να παγώσουν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αλλά και να διατηρηθούν, να επιστραφούν στην κοινωνία. Και γι' αυτό απαιτείται η κατάσχεση με εγγύηση βέβαια. Οι δείκτες υγείας και τα λοιπά. Αυτά υπάρχουν ήδη. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι όλα αυτά δεν εφαρμόζονται αποκλειστικά και ιδιαιτέρως. Είπαμε με εγγυήσει και με εναρμόνιση αυτών. Καταλαβαίνω ότι ο διαχωρισμός μεταξύ τραπεζών και ανθρώπων είναι ελκυστικός. γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι τράπεζες χειρίζονται χρήματα και ζημιώνουν την κοινωνία και τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως η ανάλυση του μαφιοζικού και μαφιοζικού τύπου φαινομένων δεν δικαιολογεί αυτό το διαχωρισμό. Μπορεί να υπάρξει και αντιστροφή των ρόλων εδώ. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στο έγκλημα που να μην έχουν καμία σχέση με τις τράπεζες. Γιατί όσο περισσότερο ολοκληρώνεται η Τραπεζική Ένωση, τόσο περισσότερο πρέπει να θυμόμαστε ότι και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρξουν πιο αποτελεσματικά ενωσιακά όργανα για έλεγχο. γιατί είναι πολύ εύκολο να διαχωρίζουμε τράπεζες με ανθρώπους, από ανθρώπους. Αλλά τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Για την Ευρωπόλ και λοιπά είπαμε ήδη ότι μερικές φορές χορηγεί Λανθασμένε ή παραπλανητικές πληροφορίες χωρίς να το κάνει επίτηδες. Δεν εννοώ ότι δεν είναι υπόλογη η Ευρωπόλ εδώ στο Κοινοβούλιο. Απλώς κάνουμε μια πρόταση για τη λισαβονοποίηση και της Ευρωπόλ. Με έλεγχο και από το Ευρωπαϊκό και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχω κάνει ακροάσεις και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό που στόχευαν στη σωστή εξισορρόπηση, αλλά όλοι συμφωνούσαν ότι η πραγματική πληροφόρηση για ορισμένες εγκληματικές περιπτώσεις δεν μπορεί να χορηγείται γενικά μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις και με συγκεκριμένους όρους. Για τον κύριο Γιακολίνο τώρα. Θα σας πω κάτι προσωπικά. Αν και το θέμα αυτό ανήκει σε άλλους, όχι σε μένα. Ξέρω λίγο πολύ τι συμβαίνει στην υπηρεσία μας, αλλά δεν μπορώ εγώ να σας δώσω τις πλήρες πληροφορίες. Κύριε Νιούτον Ντάν. Η πληροφόρηση του κοινού είναι σημαντική, αλλά από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πολιτικής συνείδησης και πραγματικής έρευνας. Γιατί μπορεί να υπάρχει συνείδηση και να μην δίνεται η διαταγή για έρευνα. Είναι και θέμα συνεργασίας θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. The political discourse is there. But Καμιά φορά οι θέσεις των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου δεν επιδεικνύουν καμία συνεννόηση. Υπάρχει θέμα κακής οργάνωσης λοιπόν. Και είναι σημαντικό να συνεχιστεί η πολιτική πίεση σε όλα τα επίπεδα, από πάνω μέχρι κάτω. πρέπει να υπάρχουν συνεχώς συμβιβασμοί και δεν φτάνουν πάντα τα πράγματα μέχρι κάτω. Πληροφόρηση λοιπόν του κοινού, ναι, αλλά για συγκεκριμένα θέματα, όχι αναγκαστικά για την ουσία της κάθε υπόθεσης, γιατί υπάρχει το ευρωβαρόμετρο που δείχνει ότι το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να λυθεί μόνο σε ενωσιακό επίπεδο ή κυρίως σε ενωσιακό επίπεδο. Όχι αποκλειστικά. Αλλά αυτό που λείπει από τις καμπάνιες πληροφόρησης δεν είναι φορά την πραγματικότητα της μαφίας αλλά το ότι πολύ συχνά δίνονται μόνο εθνικές λύσεις και όχι πανενωσιακές. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η σύνδεση που λείπει. Και λείπει και διότι η αναγνώριση όλων αυτών των θεμάτων είναι πρόσφατη. Πριν από 5-6 χρόνια δεν είχαμε τέτοιες προσδοκίες γιατί δεν υπήρχε ακόμα, δεν ίσχυε η συνθήκη της Λισαβόνας ας πούμε. Είναι πρόσφατα όλα αυτά. Αφού λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ως προς όλα αυτά, πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τον οικονομικό και όχι μόνο χώρο που ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο και σε θέματα ελευθερίας και ασφάλειας. Εν τω μεταξύ βέβαια πρέπει να συνδυαστούν και άλλα, αλλά αν η πρόταση για ευρωπαϊκό FBI είναι θετική, παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές γιατί αυτή τη στιγμή η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μου επιτρέπει γιατί δεν υπάρχει πραγματικό ομοσπονδιακό επίπεδο. Πάντως υπάρχει η Ευρωπόλ. Υπάρχει δηλαδή μια νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα για κάποια πρόοδο. Ας επενδύσουμε λοιπόν στην Ευρωπόλ. Γιατί αν ζητήσουμε κάτι καινούργιο όπως την Ευρωπαϊκή FBI καταστρέφουμε αυτό που ήδη υπάρχει και προς όφελος κάποιου πράγματος που δεν υπάρχει ακόμα. Πάντα υπάρχει τρόπος εξισορρόπησης. Για την έκθεση κατά της διαφθοράς θα έπρεπε να παρατηρηθεί πρώτα ποια στάσεις υπάρχουν στην Ευρώπη, ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι τομείς ή δημόσιες προμήθειες ας πούμε και να μην πρόκειται για απλή επανάληψη όσων έχουμε ήδη πει. αλλά συνδυασμός των πεπαρατηρημένων τάσεων σε όλες τις χώρες μέλη. Θα πρόκειται για μια πρώτη προσπάθεια με κυρίως πολιτική καταρχάς σημασία. Τώρα για τη μελέτη ξέρετε εσείς τώρα ότι που συγκρίνει Καλή ιδέα είναι, καλή, καλή. Αλλά να μην δοθεί εντύπωση ότι, ότι υπερβάλλουμε και κινούμαστε όλο και πιο πολύ προς την κατεύθυνση που ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Διότι Όλοι λένε εντάξει πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και τα λοιπά, αλλά δεν τα έχουν σκεφτεί αρκετά. Οι μελέτες που κάνουμε τη αιτήση του Κοινοβουλίου από το 11 δείχνουν κατά κάποιον τρόπο ποια είναι η τάση. Υπάρχουν και συγκριτικές μελέτες, υπάρχουν αν και πρέπει να αναγνωριστούν περισσότερες. You know, the importance and the beauty of this... Αυτή είναι η σημασία της Επιτροπής σας. Ναι, είναι τμήμα της ΕΛΕΦ ΜΕΝ, αλλά μόνο αυτή μπορεί να θίξει αυτά τα προβλήματα. Μας επικρίνουν ότι δεν κάνουμε αρκετά. ως προς διώξεις τουλάχιστον και επιβολή του νόμου. Ναι, μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, αλλά γιατί να μην κάνουμε περισσότερα. Να κάνουμε περισσότερα. Να αρχίσουν όλοι μαζί να σκέφτονται ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Διρετόρα, σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Να δώσω το λόγο και πάλι στον καθηγητή Μπικό τώρα. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το ζήτημα της ενημέρωσης κοινή γνώμης, γιατί νομίζω πως είναι βασικό. Συνδέεται με τη μεταφορά που χρησιμοποιούμε για να αντιληφθούμε το ζήτημα. Παραδείγματος χάρη, αν χρησιμοποιήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, Μιλάμε για μια οργάνωση που είναι σταθερή, στρατιωτικού τύπου και περνάμε στη γεωπολιτική. Δηλαδή, το σκεπτικό πως ο εγκληματίας είναι ξένος ε, εχθρός ε, ε, εξπακούεται και λίγα λέμε. Δηλαδή, τα πράγματα μπορεί ίσως να αλλάξουν, να αντιληφθούμε πως ε, το επίπεδο της οργάνωσης είναι μικρό μέρος ε, του ζητήματος. Εάν φαίνεται κανείς ανοργάνωτος, τι δείχνει. Ότι μιλάμε για δίκτυα, ότι είναι κάτι το οποίο μετακινείται. Οπότε δεν αναπαράγεται με τα ίδια άτομα. Κάποιοι ενδιάμεση είναι εκεί κάποια στιγμή και μετά αλλάζουν. Οπότε η δομή υπάρχει, αλλά το προσωπικό ε, αλλάζει. Είναι λοιπόν μια διαφορετική αντίληψη του τι διακυβεύεται. Αφορά έτσι περισσότερο ρευστές κοινωνίες παρά ένα φρούριο. που αντιμετωπίζει ε, έναν εισβολέα. Οπότε η αντίληψη αυτή με κάποιους ενδιάμεσους νομίζω μπορεί καλύτερα να αναλύσει το πώς στην πράξη υπάρχουν ε, διαφορετικοί τύποι σοβαρού εγκλήματος. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει διαφορετικές κατηγορίες ε, σοβαρού εγκλήματος ε, που ανταποκρίνονται σε αυτό. Τώρα, για την κοινωνική ζημία. Δεν είναι για να αρνηθούμε τη σημασία της μαφίας. Απλά για να, λέμε, για να πούμε πως προσέξτε είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο γιατί υπάρχει πολλή βία αλλά δεν είναι εξορισμού το ε, σημαντικότερο. Οπότε το σημαντικότερο είναι να επανακαθορίσουμε προτεραιότητες και πόρους στο τι θέμε ε, πραγματικά να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, μίλησα για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Απόβλητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τι προσπάθειες καταβάλουμε στο επίπεδο της Ένωσης για να καταπολεμήσουμε τα απόβλητα των μεγάλων εταιριών. Ίσως όχι αρκετά. Οπότε είναι ζήτημα προσαρμογής ίσως που σχετίζεται με το τι έχει κανείς κατά νου γιατί αν ξεκινήσουμε με κάποιο σκεπτικό θα μείνουμε στο εντυπωσιακό στο σταθερό αλλά ίσως δεν αντιληφθούμε πως υπάρχουν άλλα φαινόμενα πιο σημαντικά από αυτά τα οποία μας απασχολούν για την Europol έχουν κάνει την αυτοκριτική τους παραδείγματο χάρη για την όκτα και συνεργαστήκαμε στενά μαζί τους και είπαν πως ε, ναι, εντάξει ίσως μπορεί να κολλάμε πάρα πολύ ε, στα εδαφικά και στη γεωπολιτική και τώρα πως τώρα πράγματι ναι πρέπει να έχουν περισσότερους γεωγράφους και κοινωνικού επιστήμονες για να χαρτογραφίζουν γιατί παραδείγματος χάρη και η αίσθηση της κλίμακας είναι σημαντική αν κοιτάει κανείς ένα χάρτη σε λάθος κλίμακα, υπάρχουν τεράστια βέλη σε ένα πολύ μικρό χάρτη του κόσμου. Δημιουργούμε φόβο έτσι και δεν εξηγούμε τίποτα. Αν είναι σωστή η κλίμακα, τότε έχουμε ένα χάρτη ο οποίος θα δώσει μια καλύτερη εικόνα και με το να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα θα έχουμε μια καλύτερη αντίληψη α, ε, του τι συμβαίνει. Αντίληψη σε τοπικό επίπεδο Οπότε είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει γίνει ε, μέχρι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε κύριε Μπιγκό, ευχαριστούμε και πάλι τον ε, Διευθυντή, τον κύριο Μανσερβίση. Όπως βλέπετε είναι συνεχής η ανταλλαγή πληροφοριών και για μας είναι ζωτική σημασία, δεδομένου και του μελλαντικού ρόλου και της προοπτικής αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, επόμενους ομιλητές να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Ευχαριστώ. Για το δεύτερο πάνελ, λοιπόν, έχουμε τίτλο επιχειρηματική διαφάνεια και ποινική ευθύνη των επιχειρήσεων. Θα ακούσουμε τον Ρόμπερτ Πάλμερ από το Global Witness για την ενίσχυση της εταιρική διαφάνειας ως μέσο καταπολέμησης του οργανωσμένου και οικονομικού ε, εγκλήματος. Και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Μικέλε Ρικάρντιν, ε, ο οποίος είναι project manager της Bownet ε, του Πανεπιστημίου Transcreamer. Ο κύριος Μπίλιοντεν Μπαν, δεν ήθελα να σας διακόψω τη διάρκεια της ανακοίνωσής σας, διαδικαστικά μόνο. Πολλά μέλη του κοινού και του προσωπικού θα ήθελαν να τα ακούσουν, αλλά τους είπαν ότι όλες οι θέσεις είναι κρατημένες και δεν μπορούν να έρθουν. Από ό,τι βλέπω δεν είναι καταλημμένες όλες οι θέσεις. Ε, θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα καρτελάκια που λένε κρατημένοι για τη θέση για να μπορέσουν να έρθουν οι υπόλοιποι να ακούσουν. Δεν ξέρω για ποιον τις έχουμε κρατήσει αυτές τις θέσεις. verificando. Ναι, μισό λεπτό θα το δούμε, Μπίλ, αν υπάρχουν ε, άτομα τα οποία θέλουν να μπουν, να παρακολουθήσουν, μπορούμε κάλλιστα να τους βοηθήσουμε, να τους διευκολύνουμε. Από ό,τι μου λέει η γραμματέα όμως δεν έχει κανέναν έξω. Ok, stavo dicendo quindi il um, professore Michele Riccardi dell'Università Cattolica. Ο καθηγητής Μικέλε Ρικάρντι λοιπόν από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Τρέντο θα μας παρουσιάσει ε, την έκθεσή του για τα συμπεράσματα του Beneficial Ownership Network Project. Θα δώσω τώρα το λόγο λοιπόν στον κύριο Πάλμερ. Η συζήτηση θα γίνει ως συνήθως. Πρώτα θα δώσουμε λόγο, το λόγο λοιπόν στους ομιλητές μας, από 15 λεπτά ο καθένας και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα. Θα σας μιλήσω για την κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από άτομα που κάνουν ε, ξέπλυμα χρήματος, ε, διαφραγμένους πολιτικούς και οργανώσεις ε, του οργανωμένου εγκλήματο. Αυτό κατά την άποψή μου είναι σοβαρή αδυναμία τη καταπολέμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση του οικονομικού εγκλήματο. Θα σα εξηγήσω τι γίνεται με την ε, κρυφή ιδιοκτησία μια επιχείρηση και στη συνέχεια θα περάσω στη συστάση μου για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εγώ εργάζομαι για την Global Witness, ε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που προσπαθεί να βρει μια σχέση ε, και να σπάσει αυτό το δεσμό μεταξύ φυσικών πόρων, διαφθοράς και σειράξεων. Είμαστε πολύ γνωστοί για, την, ε, ε, ε, για το ρόλο που διαδραματίσαμε στην ρήξη για τα διαμάντια και είχαμε οριστεί για το Νόμπελ Ειρήνης. Επίσης δημιουργήσαμε την Extractive Industries Transparency Initiative, μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να ε, διαθέσει πληροφορίες για τις ε, κυβερνήσεις και τα χρήματα τα οποία προέρχονται από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και εξορυκτικές βιομηχανίες. Εγώ θα εξετάσω το ρόλο του οικονομικού τομέα και πώς το χρηματοπιτωτικό σύστημα μπορεί να ε, τροφοδοτήσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Αν είστε κλιματίας, και θέλετε να ε, κάνετε ξέπλυμα χρήματος ε, και να ε, μετακινηθείτε σε διάφορες περιπτώσεις, χρειάζεστε δύο μέσα. Καταρχάς ένα τραπεζικό οργανισμό ή κάποιον ενδιάμεσο, ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να πάρει τα χρήματά σας και να τα μεταφέρει δια ε, μέσου της τράπεζάς του. Και υπάρχει ένα πολύ καλό οργανωμένο δίκτυο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι πολύ δύσκολο στους εγκληματίες να ε, έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τρίτη οδηγία για την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εισόδων και υπάρχει και μια σχετική task force. Υπήρχε πρόσφατο το επεισόδιο με την HSBC και το πρόστιμο των 5 εκατομμυρίων δολαρίων και αυτό καταδεικνύει ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Ε, οι τράπεζες πολλές φορές παίρνουν χρήματα από διεφθαρμένους πολιτικούς οργανωμένο έγκλημα και ε, εγκληματίες. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε ένα αυστηρότερο σύστημα και συγκεκριμένες ποινές. Ε, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις ε, τράπεζες και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την συμπεριφορά των τραπεζών θα έπρεπε να φυλακίζονται. Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνονται επιτόπου έλεγχοι σε τράπεζες, να ελέγχονται λογαριασμοί και να είμαστε βέβαιοι ότι οι τράπεζες ε, κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν στην πράξη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζεται κάποιο ο οποίο θέλει να κινήσει παράνομα χρήματα είναι να βρει μια τράπεζα να μεταφέρει τα χρήματά του. Το δεύτερο το οποίο χρειάζεται είναι ένα τρόπο να κρύψει την ταυτότητά του. Αν είστε εγκληματία. <laughs> εγνωσμένου κύρους που θέλετε να μετακινήσετε χρήματα από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν χρειάζεται με το όνομά σας ε, να κάνετε λογαριασμό. Στο παρελθόν ε, πήγαιναν οι εγκληματίες με το όνομά του και άνοιγαν λογαριασμό, αλλά τώρα δεν λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι κάποιο ηλίθιος για να πάει να ανοίξει λογαριασμό, αν είναι δεφιαρμένο και κινεί παρανόμως χρήματα. Τι κάνετε, χρησιμοποιείτε μία ε, επιχείρηση βιτρίνα ή κάποια άλλη δομή για να κρύψετε την ταυτότητά σας και να κρύψετε τα εισοδήματά σας. Μία πρόσφατη έκθεση από την Παγκόσμια Τράπεζα διαπίστωσε ότι στο 77% των υποθέσεων που, ανέθεσαν, ε, που εξέτασαν συγγνώμη, ε, υπήρχε μία ε, επιχείρηση πίσω από τον ε, εγκληματία ε, που χρησιμοποιεί, εικονική η οποία χρησιμοποιούσε τα χρήματα. Σκεφτείτε το ως μία ρώσικη κούκλα με ε, Υπάρχουν διαφορετικά στρώματα και όλοι αυτοί υποκρύπτουν τον εγκληματία. Και πολλές φορές αυτά τα διαφορετικά στρώματα βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι δυνάμει τη τάξεω ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να γνωρίζει ποιο κρύβεται πίσω από μια επιχείρηση, να κατανοήσουν τι ακριβώ συμβαίνει, ποιο έχει τον έλεγχο και ποιο υποφελείται από τη δραστηριότητα τη συγκεκριμένη εταιρεία. Νομίζω ότι θα μπορούσα να σα δώσω κάποια παραδείγματα για να δείτε πώ θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, η διαφθορά, ε, είναι στην χειρότερη περίπτωση σε φορολογικούς παραδείσους, ε, στις Παρθένες Νήσιονς ε, ή στα πιο κοντινά νησιά, στο Γκέντζι, στο Τζέρζι και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εμείς πολύ συχνά στις έρευνές μας είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για τους εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν εικονικές επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μετακινούν τα χρήματά τους. Πέρσι, η Global Witness ε, δημοσίευσε μία έκθεση ε, με την ονομασία Grave Secrecy που ασχολήθηκε με ε, ένα σοβαρό περιστατικό νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων από μία τράπεζα στην Κεντρική Ασία και οι περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιήθησαν για τη μετακίνηση κονδυλίων και να υποκρύψουν την ταυτότητα του ε, εγκληματία ήταν τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, ε, ε, επιχειρήσεις συγγνώμη, του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε εικονικές επιχειρήσεις λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα μητρό μετόχων και εκεί καταγράφονται ε, ποιοι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτε μια επιχείρηση. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται κάποιο να κάνει είναι να έχει μια επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία με τη σειρά τη είναι ιδιοκτησία μια άλλη επιχείρηση σε μια άλλη ε, χώρα στην οποία δεν έχει υποχρέωση να δημοσιεύονται ε, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη τη επιχείρηση και επομένω έχουμε εικονική επιχείρηση. Και τι κάνουμε, πληρώνουμε έναν επαγγελματία για να βάλουν ε, έναν, κάποιον άλλον, ο οποίο να βάλει ένα όνομα ε, και να πει ότι αυτό είναι ο νόμιμο ιδιοκτήτη τη επιχείρηση, ενώ στην πραγματικότητα παίρνει οδηγίε από εσά που είστε εγκληματίε. Ε, άλλο παράδειγμα, πρόστιμο 185 εκατομμυρίων δολαρίων στην ε, γερμανική επιχείρηση Daimler για ε, δωροδοκία διαφόρων ανά τον κόσμο. Και τι έκαναν, χρησιμοποιούσαν εικονικές επιχειρήσεις για να πληρώνουν και να δωροδοκούν πολιτικούς. Οι εικονικές αυτές επιχειρήσεις ήταν ε, επιχειρήσεις με έδρα χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Κύπρο μεταξύ άλλων. Και τουλάχιστον σε μία περίπτωση υπήρχε ένας λογαριασμός σε μια τράπεζα στη Λετωνία ε, στο όνομα μιας εικονικής επιχείρησης. Ενώ στην πραγματικότητα ο έλεγχος ήταν ε, Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Άλλα παραδείγματα είναι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτ, ο οποίο χρησιμοποιούσε χιλιάδε κυπριακέ εικονικέ επιχειρήσει ε, για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στη Βοσνία και στο Κωσφοπέδιο και η κυβέρνηση τη Ουκρανία που χρησιμοποιεί επιχειρήσει από τη Γερμανία, τη Μάλτα και την Κύπρο για να μπορέσει να ε, γλιτώσει τι διεθνεί κυρώσει και να χρησιμοποιεί τα κονδύλια τη καταλήλω. Με άλλα λόγια, θεωρητικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ε, ε, μάλλον οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούνται μόνο στη θεωρία. Υπάρχουν απτά παραδείγματα που μας αποδεικνύουν ότι όντως χρησιμοποιούνται επιχειρήσεις με έδρα ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε ποιο είναι στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτη, ε, αυτό που ελέγχει και επωφελείται από τα κονδύλια μια επιχείρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, οι βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση συλλέγονται και δημοσιεύονται, υπάρχει το όνομα, οι διευθυντές, ακόμα και η μετοχή της. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι πληροφορίες για το άτομο που τελικώς έχει τον έλεγχο της επιχείρησης και έχει και όλα τα ωφέλη. Και αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ο τελικός δικαιούχος, ο τελικός ιδιοκτήτης και αυτός θα πρέπει να είναι ζωντανό πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι άλλη επιχείρηση. Κατά την άποψή μου, οι πολιτικοί, οι μαφιόζοι, αυτοί που φοροδιαφεύγουν, ε, οι οργανώσεις ε, της μαφίας δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εικονικές επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κρύψουν τα χρήματά τους. Η Global Witness λοιπόν πιστεύει ότι θα πρέπει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων να συλλέγουν πληροφορίες και να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και δεν είναι μεγάλη επέκταση της κυβερνητικής εξουσίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μητρό επιχειρήσεων και καταγράφει όλες αυτές τις πληροφορίες. Στην πρότασή μα, ε, μία επιχείρηση θα είναι υποχρεωμένη να υποβάλει πληροφορίες για τον ε, τελικό ιδιοκτήτη τη, όπως ε, παρέχει πληροφορίες για τους λογαριασμού της ή για τους διευθυντέ τη. Εάν αλλάξουν οι πληροφορίε του ιδιοκτήτη, τότε θα ενημερώνεται το Μητρό εντό εύλογου χρονικού διαστήματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα με 2% μόνο των επιχειρήσεων ε, που είναι καταγεγραμμένες στα Μητρό έχουν ένα περίπλοκο καθεστώς και είναι υποχρεωμένες να ε, δηλώσουν άλλο ιδιοκτήτη από τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν ε, λογικά πολύ απλές δομές. δεν είναι πολύ δαπανερία επίσης η πρότασή μας. Είναι φθηνότερο από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή και έγιναν δύο αναλύσεις κόστους ωφελία για το θέμα αυτό, μία από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2002 και μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007. Και στις δύο μελέτες κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι το να δίνονται πληροφορίες του τελικού ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης είναι φθηνότερο από το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η Global Witness ε, ε, ε, προσέλαβε ένα σύμβολο για να εξετάσει το κόστος και υπολογίστηκε ότι θα υπάρχει ένα κόστος 20 εκατομμυρίων λιρών συν έξτρα κόστος συντήρησης του Μητρώου 4 εκατομμυρίων το χρόνο. Επιπλέον, θα δαπανούνται 10 εκατομμύρια λίρε ετησίω για να διασφαλίσουμε ότι συλλέγονται αυτέ οι πληροφορίε. Αυτή τη στιγμή επαγγελματίε ενδιάμεση, τράπεζε, νομικοί, εταιρείε που παρέχουν υπηρεσίε είναι αυτέ οι οποίε είναι αρμόδιε να βρουν ποιο είναι ο τελικό ιδιοκτήτη μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιπλέον δαπάνε, διότι κάθε φορά που πάει μια επιχείρηση να ανοίξει λογαριασμό τράπεζα, πρέπει να γίνουν όλοι οι έλεγχοι από την αρχή και επίσης μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και για τις ε, αστυνομικές και δικαστικές ε, αρχές να βρούνε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης. Έχω μιλήσει με ε, άτομα από την αστυνομία που μας είπαν ότι χρειάζονται έξι μήνες για να βρούνε ποιος κρύβεται πίσω από μια επιχείρηση και όταν το βρούνε, βρούνε ποιος κρύβεται πίσω από μια επιχείρηση, διβρίσκουν ότι είναι μια δεύτερη επιχείρηση, οπότε άλλοι έξι μήνες, μετά τρίτη επιχείρηση πάλι έξι μήνες Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ δαπανηρή διαδικασία και χρονοβόρα και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ποιο κρύβεται πίσω από μια επιχείρηση που εμπλέκεται σε ε, κλιματική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κάνει αναθεώρηση των κανονισμών της ε, και της νομοθεσίας της για την καταπολέμηση του, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει μεν κάποιο ο οποίος θα πρέπει να εποπτεύει την νομοθεσία, αλλά θα μπορούσε να υψώσει τη φωνή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά αυτή τη διαδικασία. Και ε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε επινοήσει ως μία ακόμα μη κυβερνητική οργάνωση. Μα στηρίζει και ο τραπεζικός τομέας, διότι ο τραπεζικός τομέας είναι υποχρεωμένος να κάνει ελέγχους βάσει της νομοθεσίας για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων και αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο και πολύ διαπανηρό για αυτούς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να είναι θέμα ε, δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό για τις ιδιοκτήτες των εταιριών και αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο εγκληματίες θα μπορούν να κινούν χρήματα και μπορεί να αναλάβει τα ενία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάστησή σας για ερωτήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικάρντι. Thank you very much for... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παλμερίδη ανέφερε παραδείγματα για το πώς οι εγκληματίες και εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν εταιρείε για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους. Θέλω να παρουσιάσω μία σύνοψη ενό έργου που χρηματοδοτήθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και αφορούσε συγκεκριμένα αυτό το θέμα. Μιλήσαμε για τι ε, μπάμπουσκε, ε, τι ρώσικε αυτέ κούκλε, που είναι και το σήμα μα. Μάλιστα, το σήμα του έργου που κάνουμε. Θέλω να δώσω λοιπόν κάποια παραδείγματα για το πώ χρησιμοποιούν οι εγκληματίε τι ε, εταιρείε ε, και μιλάμε ειδικά για μαφιόζικες οργανώσεις. Είχαμε λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις εταιρείε που βλέπετε που έσαι ένας επιχειρηματίας στη Σικελία χάρη στο οποίο ελέγχει σχεδόν 10% του κατασκευαστικού κλάδου στην Ανατολική Σικελία. Ερευνήθηκε, αποδείχτηκε πως είχε σχέσεις με τη μαφία και οι εταιρείε τους, οι του δημεύτηκαν σχεδόν όλες. Ε, χάρη σε αυτό ένας άλλος επιχειρηματίας που είχε σχέση με την Καμόρα τη φορά αυτή στην καμπανία δηλαδή ε, έλεγχε ένα μεγάλο κομμάτι όπως είπα των κατασκευών κοντά στην Νάπολη και ολόκληρο τον κλάδο της παράνομης απόρριψης σκουπιδιών και πάλι ερευνήθηκε και δημεύτηκαν οι εταιρείε του. Οπότε η ταυτοποίηση του ποιος είναι πραγματικά πίσω από μια εταιρεία, ε, μια ύποπτη εταιρεία, είναι κρίσιμο μέτρο καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος και θέλω να υπογραμμίσω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πάλμε. Δεν μιλάμε μόνο για ξέπλημα χρήματος, αλλά για διαφθορά, φοροδιαφυγή, κρύβονται κονδύλια για δωροδοκίες και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Δεδομένης ε, της σημασίας λοιπόν του ζητήματος, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ε, είναι κρίσιμη και στο Διεθνέ επίπεδο. Σκεφτείτε παραδείγματο χάρη τον ΟΗΕ ή τη σύσταση FATF και το 2003 και το 2012 και έχει αναγνωριστεί ως πυλώνας ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, χρήματος και, θα, και στην τρίτη και στην τέταρτη σχετική οδηγία που θα υποβληθεί τις επόμενες εβδομάδες. Όμως, παρόλο το ενδιαφέρον, ε, υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και το έργο μας, ε, το Bownet, ήθελε ακριβώ να δει αυτό το ζήτημα. Αρχές είναι λοιπόν οι πρακτικές. Τι κάνουν και οι ερευνητέ και οι ενδιάμεση από την άλλη. Οικονομική και μη για να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη ύποπτης εταιρεία. Τι πληροφορίες ε, χρησιμοποιούνται, ποιες είναι οι δυνατότητες ε, χρήσης αυτών των πληροφοριών και ποια είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτό και τέλος τι χρειάζεται ε, από τις ε, διοικητικές αρχές για να βελτιώσουν τις δραστηριότητε τους και ειδικά στον αφορά τη διερεύνηση των πραγματικών ιδιοκτητών. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, το Bonet ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε έξι εταίρους, ε, πανεπιστήμια, το, το κέντρο δηλαδή έρευνας Transcrime στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, το Ευρωπαϊκό Μητρό Εταιριών ε, και από τον ιδιωτικό τομέα την Unicredit και την PricewaterhouseCoopers. Μία σειρά δραστηριοτήτων λοιπόν έλαβαν χώρα, έρευνες, ε, και ερωτηματολόγια στις ε, διοκτικές και ερευνητικές αρχές καθώς επίσης και έρευνες στα μητρώα εταιριών για το ποιο είναι ιδιοκτήτης και μέτοχος των εταιριών. Και προτείναμε κάποια νέα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και επίσης το τι σημαίνει αυτό για την πολιτική. Τώρα θα περάσω στα βασικά ευρήματα της ερευνάς μας. Πρώτα απ' όλα, όταν η ε, ερευνητές και οι ενδιάμεσοι θέλουν να δουν ποιος κρύβεται πίσω από μια εταιρεία όσον αφορά τους ε, μετόχους και τους διευθυντές. Ε, αυτά είναι τα δεδομένα που κυρίως χρησιμοποιούν, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε πρόβλημα διαθεσιμότητας. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ κρατών μελών για το ποιες πληροφορίες συλλέγουν. Κάποια κράτη-μέλη δεν συλλέγουν ακόμα αυτές τις πληροφορίες. Κατόπιν υπάρχει ένα πρόβλημα ταυτοποίησης. Δηλαδή το όνομα μετόχων και διευθυντών ε, συχνά υπάρχει, αλλά άλλες πληροφορίες, π.χ. ημερομηνία γέννησης ε, και διεύθυνση αριθμός ταυτότητας, δεν υπάρχουν. Ζητήματα ακριβίας επίσης, ε, αντισυχίες για την αξιοπιστία των πληροφοριών. Οι πληροφορίες δεν ενημερώνονται πάντα. Οπότε υπάρχει και ζήτημα του κατά πόσο είναι επίκαιρε και συχνά είναι διαθέσιμες για τις ε, για ένα τύπο τεριών είτε είναι ΕΠΕ είτε όχι, ενώ δεν είναι διαθέσιμες για ενώσεις, ε, για ιδρύματα κτλ. Οπότε, εξετάσαμε τα επιχειρηματικά μητρώα και των 27 μελών και όπως βλέπετε υπάρχει ακόμα ένα 30% των μητρώων αυτών που δεν συλλέγουν και διαθέτουν πληροφορίες για τους μετόχους. Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες των, για τα στοιχεία των διευθυντών των ευρωπαϊκών εταιριών. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης λοιπόν και οι σχετικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που είναι λιγότερο διαθέσιμες. Ε, γύρω στο 20% των πληροφοριών αυτών είναι διαθέσιμο στα επιχειρηματικά μητρώα. Αυτό μόλις είπαμε. Δηλαδή, εάν καλύπτονται ε, Εάν λοιπόν οι ανώνυμες ε, εταιρείες ε, καλύπτονται σε ποσοστό 75%, οι υπόλοιπες εταιρείες ε, δεν καλύπτονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σύμφωνα με διάφορες μελέτες για το οργανωμένο έγκλημα, ειδικά οι ε, μαφιόζικες οργανώσεις χρησιμοποιούν άλλες μορφές εταιριών που στείνονται εύκολα γιατί θέλουν να έχουν τον άμεσο έλεγχο της εταιρεία. Οπότε εταιρείε οι οποίες δεν είναι ανώνυμες αλλά είναι προσωπικές εταιρείε ε, είναι σαφώς καλύτερη λύση από μια εταιρεία με μετόχους. Δεύτερον, πηγές των δεδομένων. Τα επιχειρηματικά μητρώα εξακολουθούν να παραμένουν η πιο σημαντική πηγή για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών και αυτό, παρά το ότι υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί πάροχοι τέτοιων δεδομένων. Εγώ μέτρησα γύρω στους 150 παρόχους δεδομένων για το ποιοι είναι οι διευθυντές και οι μέτοχοι των ευρωπαϊκών εταιριών. Οπότε το θέμα δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα των ε, πληροφοριών. Πρώτον, οι περισσότεροι από αυτούς τους παρόχους και τα Μητρώα καλύπτουν μόνο μία χώρα κάθε φορά. Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των διαφορών μητρώων στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό έχει κρίσιμη σημασία γιατί όπως ε, ε, μας υπερθύμισε ο κύριος μας σερβίζει το οργανωμένο έγκλημα είναι εξορισμού διεθνές και οι διασυνοριακές έρευνες ε, είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη σημασία για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Και όταν είναι τα δεδομένα διασπαρμένα, ε, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για την έρευνα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Το πρόβλημα της ταυτοποίησης οι χρήστες ε, και τυχόν ερευνητικές αρχές και τράπεζες και επαγγελματίες έχουν πρόβλημα στο να ε, ξέρουν σε ποιο μητρό πρέπει να αναζητήσουν τα στοιχεία. Υπάρχουν τόσα πολλά και δεν ξέρουν ε, ποιο είναι αυτό το οποίο θα έχει τις πιο έγκυρες πληροφορίες. Υπάρχει και πρόβλημα πρόσβασης, ειδικά όταν μιλάμε για ξένα σε άλλη χώρα και τα περισσότερα ζητάνε πιστοτική κάρτα που συχνά δεν έχουν οι ερευνητές. Και υπάρχει και το ζήτημα του ε, κόστους. Ε, δηλαδή τα εμπορικά ε, μητρώα είναι πάρα πολύ ακριβά συνήθως και δεν μπορεί να ζητήσει κάτι τέτοιο κάποιος ο οποίος κάνει μια έρευνα. Οπότε όταν θέλει να αναζητήσει πληροφορίες ε, από ξένο μητρό συνήθως ζητά από τους ξένους ομολογούς του βοήθεια και έτσι χάνεται χρόνος και βεβαίως κοστίζει και ε, χρήμα. Και οι ενδιάμεσοι βεβαίως βασίζονται στους ε, πολίτες, στους πελάτες με και στα στοιχεία που παρέχουν, κάτι το οποίο βεβαίως όπως φαντάζεστε δεν είναι και το πιο αξιόπιστο ως πηγή πληροφοριών. Τέλος, υπάρχει η έλλειψη λογισμικού τη σήμερον ημέρα για να μπορέσουν να συλλέξουν τα δεδομένα από διάφορα μητρώα επιχειρήσεων. Οπότε δραστηριότητες όπως η ταυτοποίηση του πραγματικού ιδιοκτήτη σε μια περίπτωση στην οποία έχουμε διασυνοριακή επιχείρηση και τα λεγόμενα κινέζικα κουτιά και ε, συνδεδεμένες εταιρείες συχνά γίνεται με ε, τρόπο πρόχειρο. Και στην ερώτηση που κάναμε αν χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό και οι ερευνητές και οι διάμεσοι μας απάντησαν όχι. Συμπεράσματα λοιπόν. Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως τα μητρώα ανταποκρίνονται στις ανάγκες ε, των, ε, της νομοθεσίας περί εταιριών και όχι ε, στην νομοθεσία εξοπλήματος χρήματος. Οπότε υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα προστασίας των δεδομένων. Οπότε αν δεν είναι δυνατόν να ευθυγραμμίσουμε τη συλλογή δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό σημαίνει ε, τροποποίηση του δικαίου εταιριών, τουλάχιστον μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση της πρόσβασης στα ε, υφιστάμενα δεδομένα. Οπότε, να μην έχουμε νέα δεδομένα, να βελτιωθεί η πρόσβαση στα ήδη διαθέσιμα. Να τα συνδέσουμε δηλαδή με τρόπο καλύτερο. Ειδικά στις ε, περιπτώσεις μητρών σε άλλη χώρα. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτά. Οι διασυνδέσεις μεταξύ μητρών σε διαφορετικά κρατημέλη πρέπει να ενισχυθούν και υπάρχουν ήδη κάποιες σχετικές ε, τροπολογίες. Ανέφερα τη σχετική οδηγία. Είτε λοιπόν ε, το Ευρωπαϊκό Μητρό Επιχειρήσεων ε, είτε το Μητρό Eurogroup πρέπει να ενισχυθούν. Για να μην ανακαλύπτουν κάθε φορά τον τροχό μπορούν να υπάρξουν συνδέσεις μεταξύ των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και αυτό ισχύει και για τα μητρό επιχειρήσεων αλλά και για άλλες βάσεις ε, δεδομένων. Π.χ. για το ποιοι είναι κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών ή ποια είναι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νέα συστήματα για να βοηθούν οι ερευνητέ και οι ενδιάμεσοι που θα πρέπει βεβαίω να χρηματοδοτηθούν. Και τέλος θα πρέπει να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών όσον αφορά εταιρείε, οι οποίε δεν είναι ε, ΑΕ ή ιδρύματα ή ενώσει, ε, συνδέσμους. Όλα αυτά τα δεδομένα βεβαίω πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ζήτημα τη ε, ιδιωτικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, καθηγητή Ρικάρντι. Να ξεκινήσει η συζήτηση και να δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Νιούτον Τάν. παρακαλώ. Σύντομα. Στον κύριο από το Global Witness. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, αλλά μιλούσατε για διαφθαρμένους πολιτικούς. Εμείς στην Επιτροπή μας ε, έχουμε πολιτικούς που δεν είναι διεφθαρμένοι και θέλουν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Δεν θα μπορούσατε λοιπόν να διαχωρίσετε λίγο τους πολιτικούς από τους διεφθαρμένους λέγοντας μερική πολιτική είναι διεφθαρμένη. Γιατί νομίζω αυτό ενόχλησε πολλούς συναδέλφους εδώ. Δεύτερο και σημαντικότερο, ε, αυτό που χρειαζόμαστε στην Επιτροπή μας τελικά είναι ρεαλιστικές συστάσεις, δράσεις τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να κάνετε ορισμένες συστάσεις εκ μέρους του Global Witness. Τι να κάνουμε στο μέλλον δηλαδή. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Γιακολίνο. Ναι, Άκουσα και εγώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δύο παρεμβάσεις και τις εκτιμώ ιδιαίτερως. Να περάσω απευθείας την ερώτηση ή μάλλον τις ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω και στους δύο. Το θέμα είναι να βρούμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις ε, παράνομες δραστηριότητες. Και βεβαίως η σχέση με τα όσα συζητούσαμε προηγουμένως είναι η ποιότητα και η επιλογή των διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αναφερθήκαμε και στην τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που είναι εν εξελίξη και τη συζητάει η αρμόδια Επιτροπή για την Εσωτερική Αγοράς. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το ε, πλαίσιο και έχετε εξετάσει το κείμενο. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θεωρείτε εσείς ότι είναι χρήσιμα και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο στάδιο των τροποποιήσεων ε, που θα συζητήσει το Κοινοβούλιο πριν εγκρίνει την έκθεση. Υπάρχουν δυνατότητες αυτορύθμισης μεταξύ τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων και επίσης σε ποιο βαθμό υπάρχει σχέση μεταξύ των πληροφοριών που θα έπρεπε να λαμβάνονται προκειμένου να επιτευθούν οι στόχοι μας και το θέμα της προστασίας δεδομένων ε, και της ε, προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε και τις δύο αυτές, ε, προσπαθώντας ταυτόχρονα να επιτύχουμε και τον τελικό μας στόχο, να έχουμε όλο ένα και περισσότερες και ποιοτικές πληροφορίες. αν και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι χρήσιμος ο ρόλος όπως, ε, οργανώσεων όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια ε, για την πρόληψη και την προστασία από αυτά τα φαινόμενα και τέλος όσον αφορά το θέμα της νομικής ε, ποινής για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να βρούμε και ποινικού τρόπου δίωξη και στα κράτη-μέλη στα οποία ακόμα δεν προβλέπεται το θέμα αυτό. Θεωρείται λοιπόν ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι ε, λογική για τα όσα συζητάμε και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχει σχέση με τα όσα συζητούμε το ε, να υπάρχει το αδίκημα της ε, αυτοανακύκλωσης, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που κάνει ο ίδιος ε, ο δράστης. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βέβαια πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν σε εταιρείε γιατί και εγώ τέτοιο είμαι μέτοχος. Επομένως, αν όχι εναρμόνιση, τουλάχιστον πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους γνώση, συνεννόηση μεταξύ μετόχων και ιδιοκτητών. Μιλήσατε για εξαμηνιαίες περιόδους εσείς έξι, με την υπολογίστρια. Εγώ δεν ξέρω. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να πάρουμε μερικά μέτρα, καλό θα ήταν. Και εξισορροπημένα βέβαια. Δεν θέλουμε περισσότερη γραφειοκρατία. Πα, Ελπίζω λοιπόν να μην αυξηθεί και το κόστος με αυτά όλα. Τώρα, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας δεδομένων. Ναι, λεπτό θέμα, λεπτό. Λεπτό. Και λεπτό και λεπτό. Μήπως έχετε και γι' αυτό καμιά ιδέα. Ωραία. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ένα-δυο πράγματα. Όσον αφορά αυτή τη διαδοχική αλληλουχία έξι μηνών και άλλων έξι μηνών και έξι μηνών που προσπαθούμε να βρούμε ποιος κρύβεται πίσω από κάποια εικονική επιχείρηση, ο κύριος Σμιτ διευκρίνησε λίγο την κατάσταση στη χώρα του και μας είπε ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι γνωρίζαμε και στο παρελθόν και γνωρίζουμε και τώρα τι κάνω εγώ και τι έχω στη διάθεσή μου. Ποια είναι η ευθύνη κατά την άποψή σας και ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Διότι για μένα εκεί έγκυται το πρόβλημα. Οι χώρες μέλη είναι αυτές οι οποίες ορισμένες φορές επενδύουν ελάχιστα στο θέμα αυτό, σε συγκεκριμένες δομές. Τα κράτη-μέλη ίσως ε, κάποιες φορές ε, δεν διευκολύνουν τη ροή πληροφοριών. Τα κράτη-μέλη ίσως σε κάποιες περιπτώσεις είναι αυτά τα οποία δεν θέλουν να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και κλείνονται στο καβούκι τους. Ίσως λοιπόν η πολιτική η οποία στη συνέχεια ε, ξανατίθεται προς από ευρωπαϊκής ε, σκοπιάς είναι στην πραγματικότητα καρπός των εθνικών θέσεων. Θα έπρεπε ίσως να προσπαθήσουμε και να επιβεστητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη όχι μόνο όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους, αλλά και τις υποχρεώσεις του, τα καθήκοντά τους, διότι, επαναλαμβάνω, πολύ συχνά υπάρχει ένα φράγμα. Ζητούνται κάποιες πληροφορίες, ζητούνται μία σειρά από πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες ώστε να μην χρειαστούμε έξι μήνες αλλά μια βδομάδα ή και λιγότερο διότι ζούμε και σε καιρούς προηγμένης τεχνολογίες. Μια βδομάδα πολύ είναι. Κατά την άποψή μου είναι υπερβολικό για να προσπαθήσουμε να βρούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας συγκεκριμένη επιχείρησης. Εκεί βέβαια επισερχόμαστε σε ένα άλλο πεδίο, αλλά θα έπρεπε ίσως να υπάρχει μια πιο η ισχυρή σύσταση, πιο συγκεκριμένη, διότι πολύ συχνά ακούμε γενική φύσεως συστάσεις, χρήσιμες μεν, αλλά πολύ γενικόλογε. Ε, και επειδή ο ρόλος της Επιτροπής μας ε, ε, είναι, όπως υπενθύμησε ο κύριο Μασερβίζη, είναι πολύ συγκεκριμένος. Στεκόμαστε σε πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Και υπάρχουν ένα σωρό από θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι η μητρική μας Επιτροπή. Ε, λεπτομέρειες όμως, οι οποίες ε, είναι πολύ σαφείς, είναι στοιχειώδεις για μας και γι' αυτό το επαναλαμβάνω και συχνά. Εάν θέλουμε να εναρμονίσουμε το σύστημα, θα πρέπει να περάσουμε και από αυτή τη διαδικασία. Και πάλι λοιπόν θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο. Θα απαντήσει πρώτα ο κύριος Πάλμερ και μετά ο καθηγητής Ρικάρδη. Παρακαλώ. Thank you very much for your πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν υπενόησα πως κάποιο μέρος της Επιτροπής ήταν διεφθαρμένο. Μιλάμε για μια μικρή μειοψηφία, ελπίζουμε, πολιτικών εταιριών κτλ. που μπορεί όμως να έχει φοβερό αντίκτυπο. Εγώ εστιάζω στον αναπτυσσόμενο κόσμο και βλέπουμε πάρα πολλά παραδείγματα που τα λεφτά πάνε στις τσέπες ε, των πολιτικών που τι χάνει να είναι διεφθαρμένοι και δεν εξοδεύονται μετά σε, στις υπηρεσίες που θα έπρεπε. Ε, ευχαριστώ επίσης να σας δώσω πιο λεπτομερείς ε, προτάσεις. Δεν έχω δει την ε, τελική πρόταση για την οδηγία ξεπλήματος χρήματος. Είμαστε σε επαφή με τον Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ και είπε πως θεωρεί πως το ζήτημα του κρυφού ιδιοκτήτη εταιρεία έχει κέρια σημασία και ελπίζω να το αντιμετωπίσει εντός της ε, οδηγίας. Ελπίζω λοιπόν πράγματι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του πραγματικού ιδιοκτήτη. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε είναι το θέμα της ισορροπίας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τεράστια γραφειοκρατία στην συντριπτική πλειοψηφία των νομίμων εταιριών για να επεκταθώ. Μιλάμε κυρίως για εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, γιατί υπάρχουν ήδη διατάξεις ε, σχετικές για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες. Μιλάμε για μικρότερες λοιπόν εταιρείες, ε, ανώνυμες μεν, αλλά μη εισηγμένες. Όσον αφορά τον ε, αντίκτυπο, ανάλυση που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2002 εκτιμά πως ε, μόλις 1 με 2% των εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου θα δυσκολευτούν να ε, βρουν ποιος είναι ο πραγματικός τους ε, ιδιοκτήτης. Δηλαδή, 1 με 2% των εταιριών έχουν περίπλοκη δομή που απαιτεί κάτι παραπάνω από μια απλή σκέψη. Για τις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες απλά θα τσεκάρουμε ένα κουτί και θα, θα λένε ότι ο νομικός ιδιοκτήτης είναι ιδίως με τον πραγματικό. Όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι πράγματι σοβαρές αυτές οι ενισχύες. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η σχετική βρετανική νομοθεσία δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή νομικό εμπόδιο για την συλλογή του δεδομένου αυτού του ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ήδη συλλέγουμε και δημοσιεύουμε στοιχεία για τον ε, νομικό ιδιοκτήτη και τον διευθυντή ε, των εταιριών. Λίγο παραπέρα πάμε, δεν βλέπω τεράστια εισβολή στην ιδιωτική ζωή των πολιτών ή εταιριών. Η άποψή μου είναι πως εάν θέλει κανείς ε, να έχει τα ωφέλη της περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή να μπορεί να επιχειρεί πρέπει να πληρώσει και το τίμημα, να αποκαλύπτει ποιος είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα πραγματικό λόγο, εάν είναι κάποιος ειλικρινής επιχειρηματίας να... ή ε, μια τίμια επιχείρηση να θέλει να κρύψει ποιος είναι από πίσω. Για αυτό το οποίο είπατε τώρα, κύριε Αλφανό. Όπως έχει δείξει το έργο Bonet, ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το τι πληροφορίε συλλέγονται, η ποιότητα των πληροφοριών, ποιες πληροφορίε δημοσιεύονται και νομίζω πω η Ένωση και η ε, Επιτροπή σα μπορεί να βοηθήσει με το να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών, να ασφαλίσει πως έχουμε παρόμοιε πληροφορίε, που συλλέγονται σε όλα τα κράτη-μέλη που θα χρησιμοποιούνται κατόπιν γρήγορα και, ε, και μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν Συχνά βεβαίω είναι δύσκολο να βρεθούν αυτέ τι πληροφορίες. Μίλησα για ένα εξάμεινο γιατί συχνά δεν συλλέγονται ή δεν βρίσκονται εύκολα αυτέ τι πληροφορίε ή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Αν πάμε παραδείγματος χάρη στου παραδοσιακού φορολογικού παραδείσους, δύσκολα θα δώσουν στοιχεία για το ποιο είναι πίσω από μια εταιρεία. Τα λεφτά σήμερα ημέρα κάνουν τον γύρο του κόσμου σε δευτερόλεπτα και οι διοκτικές αρχές ε, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να παρακολουθήσουν αυτή την πορεία και να δουν ποιο κρύβεται πίσω από μια εταιρεία. Οπότε, όπω είπα στην αρχή, ευχαρίστω να σα κάνω πιο λεπτομερεί συστάσει και σχόλια για το σχέδιο οδηγία όταν θα το δημοσιεύσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ, κύριο καθηγητή. Αν δεν σα πειράζει, θα απαντήσω στα Ιταλικά. Λοιπόν, το κείμενο τη τέταρτη οδηγία δυστυχώς ε, δεν έχουμε καταφέρει να το αναλύσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποιες υποθέσεις επί τη βάση συστάσεων του ΦΑΤΦ που είναι συστηματικά το κριτήριο βάσει του οποίου αναθεωρούνται οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτός ο νέος πιο σημαντικός ρόλος για τα μητρέα επιχειρήσεων και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις ε, και στις συστάσεις του ΦΑΤΦ, διότι τα μητρώα αυτά και οι επιχειρήσεις είναι αυτά τα οποία θα διατηρούν και θα μπορούν να διαθέσουν ε, ένα σύνολο ελάχιστων πληροφοριών για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιοι είναι οι μέτοχοι μιας επιχείρησης, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ε, ερευνητές και ενδιάμεση σε πολύ γενικό επίπεδο αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι έχουμε μία βαθμιδόν ε, αλλαγή από το ρόλο των ενδιαμέσων που είχαμε στην τρίτη οδηγία κατά της νομοποίησης παρανόμων εσόδων σε μία προσέγγιση όπου και τα μητρώα πλέον και επιχειρήσεις ε, καλύπτουν ε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, δυνατότητε τη αυτορύθμιση μεταξύ των ενδιαμέσων ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Από κωδικού και δυνατότητε τη αυτορύθμιση ε, έχουμε μπουχτίσει. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και στην Ιταλία και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε αντίστοιχα πράγματα. Και δεδομένε λοιπόν αυτή τη νέα φύση και αυτού του νέου ρόλου των μητρών των επιχειρήσεων, αυτοί οι κώδικε αυτορύθμιση ε, ελπίζω να οδηγήσουν σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μητρών επιχειρήσεων και των ενδιαμέσων και των ε, ερευνητών ή ανακριτών που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες ε, που περιλαμβάνονται στα μητρώα. Τώρα, το κατά πόσο αντίθεται θέμα ε, προστασίας δεδομένων και παραβίασής τους. Εγώ δίνω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Οι προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν στην παρουσίασή μου προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Δεν θέλουμε να δημιουργηθούν και να συλλεχθούν νέες πληροφορίες. Αυτό που προτείνουμε είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες δημοσίως. Αν δείτε το διάγραμμα εδώ, διαπιστώνετε ότι πολλές πληροφορίες, για παράδειγμα για τους μετόχους, είναι δημόσιες πληροφορίες, πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να συλλεχθούν από οποιοδήποτε χρήστη. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι να οργανωθούν καλύτερα αυτές οι πληροφορίες, ιδίως όταν πρέπει να κάνουμε συσχετισμό μεταξύ διαφορετικών μητρών επιχειρήσεων. Τώρα, στις πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, αυτά τα συστήματα με τη, ε, τα ρόσκα κουτιά, τις μπάμπουσκες, ε, που υπάρχουν επιχειρήσεις που κρύβονται πίσω από άλλες επιχειρήσεις, αυτό που χρειάζεται ως στοιχείο της διαδικασίας ανάκρισης είναι να βρούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα μητρώα μεταξύ των και νομίζω ότι έχουμε υπερεκτιμήσει λίγο το χρόνο που χρειαζόμαστε για να βρούμε ποιο είναι ο πραγματικό ιδιοκτήτη ε, μια σειρά εικονικών επιχειρήσεων και για να μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίε για το ποιο είναι αυτό ο οποίο στην πραγματικότητα επιφελείται από τα κονδύλια αυτά. Μπορεί βέβαια 6 μήνε να είναι πάρα πολύ, ε, αλλά πρόκειται για πληροφορίε, οι οποίε αυτή τη στιγμή δεν μα είναι διαθέσιμε απευθεία. Επί παραδείγματι, εδώ έχουμε αυτό το διάγραμμα, ε, τα δύο διαγράμματα που σας έδειξα στην παρουσίασή μου των ε, ε, ιδιοκτητών που βρίσκονται και εδρεύουν στην Ιταλία. Και αυτά τα δημιουργήσαμε βάσει πληροφοριών που λάμβαναν σε ένα μητρό επιχειρήσεων μέσα σε μια εβδομάδα. Στις περιπτώσεις τις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές έδρες σε άλλες χώρες, ε, για να μπορέσουμε να, κάνουμε, να ανατρέξουμε στο σύστημα και να βρούμε ποιος είναι ο τελικός ιδιοκτήτης, τότε σίγουρα μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση. Infine, ruolo ε, delle Τέλος, ο ρόλος των εμπειρικών επιμελητηρίων, ε, όπως υπενθύμησα και στην αρχή, είναι ζωτική σημασίας, ολοένα και περισσότερο μάλιστα, και αυτή τη στιγμή αναγνωρίζεται και από τα ίδια τα εμπορικά επιμελητήρια ε, ο ρόλος αυτός και υπάρχουν και διάφορα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των οποίων τα εμπορικά επιμελητήρια ε, δραματίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να προτείνουν ε, και λογισμικό αλλά και κάποιες πλατφόρμες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για να γίνονται έρευνες για τα θέματα του ποιος είναι ο τελικός ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, διακόπτουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα και να σας υπενθυμίσω ότι από τις 5.30 έως τις 6.30 θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και περιμένουμε να μας δώσετε και τη γραπτή σας συνεισφορά. Καλό μεσημέρι.